Θα δώσω τώρα το λόγο στην συνάδελφο Χέντζερ. Ευχαριστώ ναι. πολύ και σας ευχαριστώ για όλες τις συμβολές σας. Πιστεύω πως ακούστηκαν πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες και είμαστε και οι δύο ευγνώμονες για την συμβολή σας όσον αφορά τα περαιτέρω βήματα που ελπίζουμε ότι θα χρειαστεί να κάνουμε με τη δική μας έκθεση. Η ιδέα δηλαδή ότι χρειάζεται να επιμένουμε και στην διαβίου μάθηση είναι πολύ σημαντική και πρέπει όντως να συμπεριληφθεί σε επόμενες ε, μελέτες για την ενεργειακή κοινότητα. Να στραφώ στα τρία ερωτήματα που έθιξε ο κύριος Τούρμες ας πούμε, για την εισαγωγή μιας ιεραρχίας όπως έχουμε στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Είναι Πολύ τιμό το σχολείο σας και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη ειδικά εάν θέλουμε να συνδυάσουμε την ε, κεντροποίηση και την αποκέντρωση. Ε, γιατί χρειάζεται η ιεραρχία κανόνων για να κατευθύνει τις αποκεντρωμένες ενέργειες. Εμείς ε, δεν έχουμε δόγματα. Εδώ έχουμε μιλήσει μόνο για την συνθήκη άνθρακα και χάλιβα μια νομολογία όπου υπάρχει εκεί όσον αφορά την προειδοποίηση για την υπερβολική απόδοση ε, αρμοδιοτήτων σε εκτελεστικές, ε, εκτελεστικούς οργανισμούς. Αυτό ελήφθη υπόψη πολύ σοβαρά και ερμηνεύθηκε έτσι στις, ε, στην εντολή λειτουργίας του Acer. Η Λισαβόνα μπορεί να μας προσφέρει ε, βέβαια το πλονέκτημα του να απομακρυνθούμε από τις πολιτικές ε, και νομικές δεσμεύσεις του περίφημου, της περίφημης Μαρόνι. τελευταία ερώτηση αφορούσε το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την μόχλευση με την αγορά φυσικού αερίου. Αν μπορούμε δηλαδή να έχουμε ε, πιθανές ρυθμίσεις για την αγορά φυσικού αερίου. Όντως εκεί θα ήταν καλό το να παρουσιάσουμε μια, ένα πιο συμπαγές μέτωπο, να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε και την αλληλεγγύη ως αγοραστές. Όπως ανέφερα, χωρίς να παραβαίνουμε τους κανόνες αντιτράστ, αλλά έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο βάρος Ίσως αυτό θα μπορούσε να γίνει δυνατό μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών με ανάμεσα στις εταιρείε, διαπραγματεύσεις με έναν μόνο προμηθευτή, που να προσπαθήσουμε να έχουμε δηλαδή μια κοινή πλατφόρμα. Αλλά φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να δουλευτούν περισσότερο και να έχουμε ε, και περισσότερες ιδέες για το πώς θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις επεξηγήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Και Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν σύντομε ερωτήσει. μπλε κάρτε. Ναι, δύο έχω, έχω ερωτήσει, ίσως όχι παραπάνω από τρει-τέσσερι. Τριάντα δευτερόλεπτα για ερωτήσει. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, είμαι Βέλγος και μέλος της Επιτροπής Περιφερειών. Θέλω να σας συγχαρώ για την οργάνωση αυτής της ημερίδας και να ευχαριστήσω τους δύο εμπειρογνώμονες. Συμφωνώ με τη γνώμη τους ότι η Ευρώπη χρειάζεται νέα πνοή. Πιστεύω ότι μία ε, νέα συνθήκη ενεργειακή θα δώσουν αυτή τη νέα πνοή. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να ε, ε, ονειρευόμαστε αλλά να βρούμε και μία μέση οδό διότι η κοινότητα αυτή θα επιτύχει μόνο εάν συμφωνήσουν ε, οι κοινότητες μας και η τοπική αυτοδιοίκηση θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό και η συμφωνία των δημάρχων που έχει προωθήσει η Επιτροπή των Περιφερειών είναι ε, μία βασική κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση και οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο και να αξιοποιήσουν τη συμμετοχή του πληθυσμού μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση και ερώτησή σας για το θέμα αυτό. Ο κύριος Σφόμποντα, πολύ σύντομα προς τους συντάξαντες τη μελέτη. Είμαι εδώ. Ίσως κάνατε τη μελέτη. Ε, τι θα γίνει τώρα, δηλαδή ε, πώς θα προχωρήσετε ως προς τις λεπτομέρειες, θα ακολουθήσετε τις ιδέες που θα παρουσιαστούν εδώ, διότι θα πρέπει να προχωρήσετε. Ποιες είναι οι λεπτομέρειες, ποια είναι, η... ποια τα εμπόδια, δηλαδή εμείς τι μπορούμε να κάνουμε να αξιοποιήσουμε την μελότησή σας. Άννα Ζαρεύσκα. Ε, πολωνικά. Ευχαριστώ αυτή ε, ε, η συνεδρία είναι πολύ σημαντική αλλά πολύ σύντομα προς την ομάδα εργασίας όταν μιλάμε ε, ε, για μέτρα για να προωθήσουμε την κοινή ενεργειακή πολιτική, ο όρος ε, συνθήκη είναι σημαντικός. Θα έπρεπε να τον αποφύγουμε διότι όλοι προσπαθούν να αποφύγουν κάτι τέτοιο. Όλοι όμως επιζητούμε και θέλουμε να γνωρίζουμε καλύτερα σε τι πλαίσιο θα μιλήσουμε για μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Νομίζω ότι η πολιτική για το 2020 Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι η απάντηση και εδώ θα έπρεπε να υπάρξει η εμπλοκή μας. Τελευταία ερώτηση, σύντομα παρακαλώ. Με... Από την Εθνική, Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Λοιπόν, Όποιο λέει και ηγεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε τελικά στη γαλλική θέση και εγώ ήμουν πάρα πολύ, ενδιαφέρθηκα πολύ από τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ στα ποσοστά τη μειώσεω των αερίων θερμοκηπίου στο πακέτο κλίμα και ενεργεια 2020 2020-2020 και το ότι κάποιες λεπτομέρειες που θέλετε, δηλαδή μείωση 30-20% θα πρέπει να είναι κάτι που να ε, εξεταστεί και να θα πρέπει οι διεθνείς προσπάθειες να υπόκειται σε μια ρεσιμότητα. Όπως μιλήσαμε, χρειάζεται και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και διεθνή αλληλεγγύη. 30% πέρα από το 20%. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα μπορούσατε να προβείτε σε κάποια σύντομα σχόλια, να δώσετε κάποιε απαντήσεις στις ερωτήσεις, η κυρία Πρώτα. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Η μελέτη πώς θα προχωρήσει. Σαν πανεπιστημιακή και νομική θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να θαρρύνουμε τη συζήτηση κυρίως μεταξύ των συναδέλφων νομικών και πανεπιστημιακών που ενδιαφέρονται για το θέμα. Ξεκινήσαμε ήδη. Ε, νομίζω ότι υπάρχει και κάποιο πρόγραμμα που έχει ετοιμαστεί ε, σχετικά με την ενθάρρυνση της συζητήσεως του θέματος. Βασική μας ιδέα ποια είναι. Συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων. Για να αναπτυχθεί περισσότερο η ιδέα αυτή είναι κάτι αναγκαίο και αυτή η συζήτηση θα πρέπει να λάβει χώρα, κατά την άποψή μας, σε όλα τα επίπεδα που είναι δυνατόν. Διότι η αποδοτική χρήση της ενέργειας, η χρήση της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Και χρειαζόμαστε και την άποψη σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό και εθνικό. Είναι ζωτική σημασία. Αυτά μπορούμε να πούμε για το πώς μπορεί να προχωρήσει το όλο θέμα. Ε, δεν είναι ιδιοκτησία μας αυτή η ιδέα, δεν διατηνόμαστε κάτι τέτοιο. Αντιθέτω, ελπίζουμε όλοι να την εστερνιστούν και να την ε, συζητήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο σχόλιο όσον αφορά τη λέξη συνθήκη. Αν δημιουργεί προβλήματα στα κράτη-μέλη θα μπορούσαμε να δώσουμε άλλη ονομασία. Όπως ενιαία πράξη. Ήταν πολύ επιτυχής συνθήκη αυτή και δεν είχε αποκληθεί συνθήκη. Μπορούμε να την ονομάσουμε πράξη. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Να σας ευχαριστήσω εκ νέου, ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονές μας που παρουσίασαν τις απόψεις τους, που απάντησαν σε ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας ζητήσω να με ακούσετε για άλλα δύο λεπτά, διότι έχω σημαντικότητες πληροφορίες να σας δώσω στα πολωνικά. Λοιπόν, θα χωριστούμε σε τρεις ομάδες εργασίας. Η πρώτη ομάδα εργασίας έχει τον τίτλο «Ασφάλεια ενέργειας, ποικιλομορφία, αλληλεγγύη και αλληλεξάρτηση στον εφοδιασμό ενέργειας». Πρόεδροι, ο κύριος Χάνες Σβόμποντα, Ευρωβουλευτής, και η κυρία Σεσίλια Τόφμπουντ από τη Βουλή της Σουηδίας. Εισηγητής ο κ. Σαρουσβόσκη, ο συνάδελφός μας Ευρωβουλευτής. Αυτή η ομάδα εργασίας τα συνεδριάσει εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Η ομάδα εργασία 2 με τίτλο ε, Ενή αγορά ενέργειας, ανταγωνισμό, ρύθμιση και τιμολόγηση της ενέργειας. Συμπρόεδροι, ο κύριος Γεγέρμο Μαρισκάλ Ανάγια από το Ισπανικό Κοινοβούλιο και η κυρία Αντίνα Ιωάννα Βαλεάν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συγητής, ο κύριος Φέλιξ Λαβία Μαρτίνες του Ισπανικού Κοινοβουλίου. Αυτή η ομάδα εργασία, η ομάδα εργασία 2, θα συνεδριάσει στην αίθουσα 3C50. Είναι η αίθουσα που είναι ακριβώ απέναντι από εδώ, όταν αποχωρήσετε από την αίθουσα Ολομέλεια. 3C50, στον ίδιο όροφο. Η τρίτη ομάδα εργασία με τίτλο Ενέργεια και Περιβάλλον, Νέα Ενέργεια, Ανανεώσιμε Πηγέ Ενέργεια και Τεχνολογία. Συμπρόεδρη ο κύριο Κλοντ Τούρμε, που είναι Ευρωβουλευτή και ο κύριος Χωσέ Ιγνάθιο Παλάθιο Σουάστη από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Η εισηγητής, ο κύριος Χεσούς Αλίκουε Λόπες και εκείνο από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Αυτή η ομάδα εργασία, η ομάδα εργασία 3, θα συνεδριάσει στην αίθουσα 1α002. 1α002. Δύο ορόφου πιο κάτω από εδώ είναι ακριβώ από κάτω από αυτή την αίθουσα. Δύο και ο κάτω, ακριβώς από κάτω όμως, αυτή τη θέση. Για να πάτε στι αίθουσε για τις ομάδες εργασία. Ε, θα δείτε, έχει επιγραφές για να σας δείξουν πώ θα πάτε στι άλλες αίθουσε. Έχει πινακίδες. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τους εισηγητές να συντάξουν τις εκθέσεις τους μέχρι αύριο το πρωί στις 9, ούτως ώστε να παρουσιαστούν στην Ολομέλεια που θα διεξαχθεί αύριο το πρωί. Φοβάμαι λοιπόν ότι οι συγητές μας έχουν δουλειά για το σπίτι απόψε. Στις 7.30 απόψε θα έχουμε ένα κόκτέιλ και ανεπίσημο δείπνο. Σας καλώ όλους στο κόκτέιλ και στο δείπνο. Θα λάβουν χώρα αυτά σε αυτό το κτίριο στην αίθουσα Γεχούντι Μενουχίν, στον χώρο Γεχούντι Μενοχήν, στον πρώτο όροφο, αρκετά κοντά στην αίθουσα της ε, ομάδας εργασίας 3. Η αίθουσα λοιπόν ο χώρος Γεχούντι Μενουχίν και ξανά θα δείτε τις επιγραφές. Υπάρχουν λοιπόν πινακίδες. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί αλλά τώρα η δραστηριότητά μα είναι σε ομάδε εργασία Και μετά κοκτέιλ και δείπνο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ευχαριστώ του συνάδελφου από την Ισπανική Γερουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφα. Dear colleagues, could we start the meeting, please? On Εκ μέρους του, εκ του Συμπροέδρου, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ στην ομάδα εργασίας που δεν μπορούμε να σας δώσουμε μεγαλύτερο διάλειμμα για καφέ και τσάι. Είναι έξω. Δεν επιτρέπεται να το φέρετε το τσάι, το καφέ εδώ στην αίθουσα της Ολομέλης, στο ημικύκλιο. Είναι τιμή μου να ξεκινήσω τις εργασίες και να δώσω το λόγο στο συνάδελφο, στη συνάδελφο του Σουηδικού Κοινοβουλίου Μοχάνες Σφόμποντα. Είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1996. Είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Βιομηχανίας και Ενέργειας. Και είναι αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ασίας που σχετίζεται με τα θέματα της ενέργειας και μέλος αντιπροσωπείας για τις ΗΠΑ. Βασική ιδέα είναι εξή. Ελπίζουμε να μην επαναλάβουμε τη συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια αλλά θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή από τον εισηγητή, μετά θα γίνει σύντομη συζήτηση και στα μισά περίπου των εργασιών θα δώσω τη σκητάλη στον συμπρόεδρο ή θα πρέπει να φύγω εκτός Βρυξελών λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Να πω μερικά λόγια, απευθυνόμουν στον συγγητή, τον κύριο Σάιρος Βόλς. Ο κύριος Σάιρος Βόλς είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Πολωνία ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τότε ετοίμασε μια έκθεση για την εξωτερική πολιτική ενέργειας. Η έκθεσή μας ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα. Υπήρξε πάρα πολύ καλή συνεργασία όλων των πολιτικών ομάδων με τον κύριο Σάιος Βότσκι. η ευρεία συνένεση. Αν έχετε την καλοσύνη σας παρακαλώ λίγη ησυχία, έλεγα ότι επετεύχθη ευρεία συνένεση ε, επί των διαφόρων θεμάτων και ευρεία συνένεση όσον αφορά την πρόθεση κοινή ε, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και στον ενεργειακό τομέα. Είχαμε κακές εμπειρίες βεβαίως κατά το παρελθόν. Ίσως δεν είναι όλες οι απόψεις οι ίδιες όσον αφορά τους λόγους για τη διακοπή εφοδιασμού σε φυσικό αέριο αλλά κοινή μα θέση ήταν να μην επαναληφθεί αυτό το γεγονός και γι' αυτό το λόγο επίση, σε αυτή τη φάση προσπαθούμε να ετοιμάσουμε μια οδηγία για τον ασφαλή εφοδιασμό σε φυσικό αέριο μια οδηγία που δίνει ρόλο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει σχέδια προλήψεως μαζί με τις εθνικές κυβερνήσεις για την περίπτωση κατά την οποία θα υπήρξε ξανά διακοπή εφοδιασμού φυσικού αερίου. Εγώ είμαι σκιώδη ηγητής για την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και ελπίζουμε με πάρα πολύ καλή συνεργασία με τι πολιτικέ ομάδες να καταλήξουμε σε κάποια λύση, σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα μαζί με την Ισπανική Προεδρία. Για να σας δείξω λοιπόν ότι στις διάφορες δραστηριότητε μας κινούμεθα προσπαθώντας να κινηθούμε στο πεδίο που σκεγράφησαν οι δύο ε, φιλοξενούμενοι ε, ομιλητές που μας παρουσίασαν τη μελέτη τους. Αυτά ήθελα να πω. Τα χρονικά όρια που ίσχυσαν πριν θα πρέπει να ισχύσουν και εδώ. Θα ήθελα στην αρχή και ο Σαρσβόσκι να παρουσιάσει κάποιες βασικές ιδέες όσον αφορά το θέμα μας είναι ένας από τους εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ο Γιάτσακ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, στο Κοινοβούλιο ξεκινήσαμε τον προβληματισμό όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική για θέματα ενέργειας, όσον αφορά τον ασφαλή εφοδιασμό. Ήδη ξεκινήσαμε το 2007 και έχουμε προχωρήσει πολύ σήμερα, διότι έχουμε και τα διάφορα άθρα της συνθήκης της Ασαβώνας, κυρίως το 194. Το βασικό μήνυμα της εκθέσεως που ανέφερε ο Χάνες Σβόμποντα και είχε την καλοσύνη να την υπενθυμίσει είναι ότι θα πρέπει να μιλάμε με μια φωνή σαν ένωση και ότι θα πρέπει να κινούμεθα όλοι μαζί και θα πρέπει να αντιληφθούμε την ενέργεια όχι μόνο σαν κάτι που αφορά το εμπόριο και την οικονομία αλλά σαν κάτι που αφορά και τα θέματα ασφαλείας αφετηρία μας ποια είναι ότι από το 2006 καταλάβαμε ότι η αγορά δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην κρίση, απέτυχε. Και τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην κρίση, απέτυχαν. Και θέλουμε να βρούμε κοινοτική λύση. Για αυτό το σκοπό θέλαμε λύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως και συμπεράναμε ότι είχε καθήκον η Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει ασφάλεια σε όλα τα μέλη της και σε όλους τους πολίτες της. Ήταν η στιγμή που ξεκινήσαμε να θεωρούμε σαν γεωπολιτικό παράγοντα την ενέργεια. Είδαμε την πλήρη γεωπολιτική της διάσταση και στείλαμε ένα μήνυμα ότι χρειαζόμαστε δηλαδή πλήρη πολιτική για την ασφάλεια της ενεργείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω και είχαμε μετά και τη μελέτη Jacques Delors που υπευλήθη στη διασκεψή μα, που επεκτάθη περισσότερο στο θέμα. Η πρόκλησή μα ποια είναι όταν θέλουμε να δούμε κατά πόσο υπάρχει πολιτική βούληση και η δυνατότητα για αυτή την αλληλεγγύη, πώ να συμφιλιώσουμε την ένταση που δημιουργείται λόγω ελληνιακών πολιτικών, εκεί που χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αλληλεγγύη, και τα κράτη-μέλη θέλουν να δημιουργήσουν δικές τους δομές εφοδιασμού ταυτόχρονα. Αυτά τα δύο, πώς θα τα συμφιλιώσουμε. Και το δικό τους ενεργειακό μείγμα. Το να συμφιλειωθούν οι δύο αποκλίνουσες προσεγγίσεις χρειάζονται δύο προαπαιτούμενα. Χρειάζεται πολιτικό όραμα και βούληση και το λέω μα είμαστε μεταξύ, θε, μεταξύ θέσεως του Κοινοβουλίου και θέσεω των χωρών στο Συμβούλιο βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κοινό όραμα και βούληση, υπάρχει έλλειψη και χρειαζόμαστε και τα νομοθετικά μέσα τα οποία προετοιμάζονται και αλλάζονται και τροποποιούνται από το Κοινοβούλιο. Η οδηγία για το φυσικό αέριο, στην οποία αναφέρομαι, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ολοκληρώθηκε στο Κοινοβούλιο, την χάνει πλήρους υποστηρίξους, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία και κατεφημισμών το λέω αυτό με το Συμβούλιο και τώρα έρχεται η ώρα της αλήθειας. Θέλουμε να δούμε και κατά πόσο αξίζει και το άρθρο της 194 ε, της της Αβώνας και το σχέδιο νομοθεσίας θα αποδείξει ότι μπορούμε να μεταμορφώσουμε, να το μεταφράσουμε αυτό σε νομοθετικές πράξεις. Δηλαδή την αρχή της αλληλεγγύης και του ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού. Τα νομικά μέσα προτείνονται στην ε, νομοθετική αυτή πράξη. Κάποια μέσα αναφέρονται σε προληπτικά μέτρα, ξεκινώντας από τον έλεγχο και την αντίδραση, αν προκύψει ανάγκη, κρίση, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν, να μεταφέρονται προνόμια από επίπεδο κρατών μέρου σε κοινοτικό επίπεδο σε περίπτωση ανάγκης και θα πρέπει να το δικαίωμα παρέμβαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υπάρχει μαζική διακοπή εφοδιασμού ενέργειας και όχι μόνο όταν υπάρχει απειλή, όχι μόνο όταν συμβαίνει μάλλον, αλλά όταν υπάρχει απειλή η διακοπή του εφοδιασμού. Θέση μα είναι επίσης ότι χρειάζεται περαιτέρω κοινοτική δράση για, να, για επενδύσεις σε κρίσιμες ε, υποδομές, διασυνδέσεις κυρίως με τα συστήματα των κρατών μελών και θεσμικά προτείνουμε ο νέος φορέας μάλλον ο είπα, η ύπατη εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Ενώση, η Υπουργό Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Λέβη Άστον, θα πρέπει να έχει τι δέουσε αρμοδιότητε και καθήκοντα. Να μπορεί να αντιδρά εναντί των χωρών παροχή παροχής ενέργειας ή ε, διαμετακόμισης ενέργειας. Και κυρίως όταν συζητούνται και διαπραγματευόμεθα συμφωνίες με αυτές τις χώρες. Όλες αυτές οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν την πρόταση α, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των διαφόρων χωρών. Το όραμά μας είναι φιλόδοξο, το δέχομαι, αλλά έχουμε ισχυρή, ισχυρή αντίδραση κάποιων κρατών μελών που δεν θέλω να αναφέρω, προτιμούν να εξασφαλίσουν σε διμερές επίπεδο τον εφοδιασμό παρά να εκχωρήσουν ε, κυριαρχία και να κινηθούν μέσω κοινή δράσεως. Και το μεγάλο ερώτημα και η δοκιμή θα είναι πόσο αποφασιστικά προνόμια θα δοθούν δυνάμει το άρθρο 104 στην κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίως μέσω του νέου κανονισμού. Δεν μιλούμε ακριβώς την ίδια γλώσσα όπως η γλώσσα που χρησιμοποιεί έκθεση Delors, αλλά δεν αποκλείεται η δημιουργία κοινών ομάδων για τον εφοδιασμό σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. και υποβάλλεται σχετικά πρόταση από τη στιγμή που θα συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη. Αν δεν καταφέρουμε να κινητικοποιηθεί ο ασφαλή εφοδιασμός ενέργεια, θα πληρώσουμε υψηλό τίμημα για, τους, για τις πηγές ενέργειας, θα πληρώσουν οι πολίτες και θα κινδυνεύσουμε να έχουμε και άλλες διακοπές εφοδιασμού, εξίσου δραματικές όπως κατά το παρελθόν. Και θα υπάρξουν ενδεχομένω και γεωπολιτικές συνέπειες όσον αφορά την έλλειψη κοινωνικής δράσης, διότι κάποιες ευάλωτες χώρες στη γειτονιά μας θα υποστούν ενεργειακές πίεσεις. Θα χρησιμοποιηθεί η ενέργεια σαν πολιτικό όπλο. Και η Ένωση θα απειληθεί και θα επηρεαστεί ίσως η εξωτερική της πολιτική. Θα πιεστεί η εξωτερική πολιτική ή θα χρησιμοποιηθεί σαν πιεστικός μοχλός η ενέργεια έναντι της ενώσεως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή, για την παρουσίαση. Πολύ σύντομη, πολύ ακριβής προτείνω ζωηρή συζήτηση. Να μην ετοιμάσουμε καταλόγους κλπ. Σηκώστε το χέρι. Θα προσπαθήσω να δω το όνομά σας, δεν είναι εύκολο. Θα προσπαθήσουμε αυτό να κάνουμε όμως. Θα ξεκινήσω. Κύριο Βι... Βικάρη από την Ιταλία. Η κυρία Βικάρη από την Ιταλία θα είναι η πρώτη που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η τα ΛΙΑΝ είσαι σημαντικά τα τελευταία χρόνια της παρεμβάσεις για την εξασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας σε συντονισμό με άλλους ευρωπαίους εταίρους οι δράσεις μας έχουν σαν στόχο να ενισχύσουμε τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και να δημιουργήσουμε νέο δυναμικό δυνατότητα αποθήκευσης, να αυξήσουμε την παραγωγή της ενέργειας, να ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μαζί με επαναπροώθηση της ε, πυρηνικής ενέργειας και να χρησιμοποιήσουμε τους φυσικούς πόρους που βρίσκονται στο επέδαφος της χώρας μας. Η τελική νομοθεσία κινείται προς την απλούστευση τις ε, δυνατότητες αδειοδότησης για την υλοποίηση νέων υποδομών ενεργειακών που θεωρούνται στρατηγική σημασία για την χώρα και σχετικά όσον αφορά τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τη δημιουργία ε, διαφόρων συστημάτων ε, διανομής υγροποιημένου αερίου διπλασίασε τον τελευταίο χρόνο την παραγωγή τη Ιταλία από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και στη διαδρομή για να ξεκινήσει ξανά η παραγωγή από πυρηνικού σταθμού για να μειωθεί η εξάρτησή τη από τα ορυκτά καύσιμα και να ευθυγραμμιστεί με τι άλλε χώρε Ευρω... των G8 όσον αφορά αυτό το θέμα. Τέλο, προχωρά προ απλούστευση η Ιταλία των αδειοδοτικών διαδικασιών διαδικασιότητες εξόριξη υδρογονανθράκων, ε, όπου είναι πλούσια η Ιταλία γι' αυτό συμμορφούμενοι με, τα, με τις στον αφορά το περιβάλλον. Λοιπόν, οι προσπάθειε τίθενται στην ε, εθνική ενεργειακή στρατηγική. Ε, και η Διεθνή ε, Υπηρεσία Ενέργεια ενέκρινε τα μέτρα τη Ιταλία. Η ενεργική πολιτική μα περνά μέσα από την χρήση μέχρι το 2020 25% τη ενεργειακή πολιτική, ενεργειακή παραγωγή Αμέσω τη πυρηνική ημέρα είμαστε 0,25% από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Σήμερα είμαστε στο 8,9% και 50% παραγωγή από ρηκτά καύσιμα. Σήμερα καταναλώνουμε το 85% από εκεί. Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, αν του πετύχουμε αυτούς του στόχους, θα έχουμε μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια στη χώρα μα, αλλά όσον αφορά την αλληλεγγύη, την ενεργειακή και την ανάληψη των ευθυνών, μας έναντι των άλλων εταίρων μας των Ευρωπαίων. Μας βοηθά να, να πετύχουμε τους στόχους. Αυτή η πολιτική που ακολουθούμε. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Παλτσίτης είναι ο επόμενος. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα και στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσω τις ευχαριστίες. Ευχαριστίες ε, διότι καταβλήθηκαν προσπάθειες την ενεργειακή πολιτική να την οδηγήσουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έγιναν κάποια βήματα, προτεραιότητες θεσπίστηκαν, το πακέτο των ενεργειακών μέτρων υιοθετήθηκε και τα λοιπά. Ξέρουμε όμως πολύ καλά δεν έχουμε μια ενιαία εσωτερική αγορά για τα ενεργειακά προϊόντα. Και αυτό κυρίως για δύο λόγους. Όσον αφορά μια, την εσωτερική πτυχή, την εσωτερική συνιστόσα, φταίει, είναι η σημερινή κατάσταση. Τα κράτη-μέλη αυτό που κάνουν είναι ότι δεν υλοποιούν στο πλήρες μέτρο τις πολιτικές τους ή με τον καλύτερο τρόπο και διαφοροποιούνται κιόλας και τα συμφέροντα των κρατών μελών στα ενεργειακά θέματα και κάτι τέτοιο δεν είναι θετικό για την ενιαία ενεργειακή αγορά. Το άλλο όμω σημείο είναι η απουσία υποδομών. Δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια ενιαία εσωτερική αγορά όταν δεν υπάρχει δίκτυο υποδομών που να συνδέει τη μία χώρα με την άλλη. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια κοινή θέση όσον αφορά τους ε, ε, παρόχους των ενεργειακών προϊόντων εκ των έξω από τους οποίους εξαρτώμαστε. Και πρέπει εδώ την κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να την ξανασυζητήσουμε. Τότε Πολλά κράτη-μέλη είχαν πληγεί άμεσα. Την εξάρτησή μας από τους εξωτερικούς παρόχους πρέπει να την μειώσουμε. Πρέπει να προωθήσουμε τις υποδομές μας και να δράσουμε θετικά. Και πιστεύω ότι το δυνατόν πιο γοργά θα πρέπει να έχουμε μια ομάδα χωρών, ευρωπαϊκών χωρών, για τους αγωγούς, ώστε συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών χωρών να τα προασπίσουμε και να τα προαγάγουμε. Αυτό θα βοηθούσε στο μέλλον να αποφύγουμε τέτοιου είδους προβληματικές καταστάσεις στο μέλλον. Κράτη-μέλη, ακόμα και όταν βρίσκονται πολύ κοντά σε εξωτερικούς παρόχους, <clears throat> να μην είναι υποχρεωμένα να πληρώνουν ένα τρίτο της τιμής με περισσότερο από ότι άλλοι. Αυτό αντιβαίνει την αρχή και την ιδέα της ευρωπαϊκής κοινότητας. Και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη τα συμφέροντα όλων μας και της ενωσής μας στα ενεργειακά θέματα όταν κάνουμε λόγο για τη μελλοντική ενεργειακή πολιτική. Θα πρέπει τα συμφέροντα των 27 κρατών μελών να προαχθούν και να υπερασπιστούμε αυτά ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήταν σύντομοι οι πρώτοι ομιλητές. Και τώρα προχωρούμε. Um, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα αυτή και παρότι δεν είμαι παίων για ενεργειακά θέματα, ήδη έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Ίσως πρώτα να κάνω ένα σχόλιο για το άρθρο 194 της συνθήκης διότι βλέποντας αυτό το άρθρο συνειδητοποιεί κανείς ότι όπως και άλλα άρθρα της συνθήκης είναι ένα είδος συμβιβασμού και αυτό. Διότι στο 194.1 αναφέρονται κοινέ επιμερισμένες αρμοδιότητες ε, όσον αφορά την ε, Ένωση ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και την προστασία του περιβάλλοντος. Όμως το 194.2 λέγει ότι η συνθήκη δεν θα πρέπει να περιορίζει τα δικαιώματα των κρατών μελών για τους όρους εκμετάλλευσης των ε, ενεργειακών πόρων. Όπως φαντάζεστε, μια και προέρχομαι από μια χώρα που όταν ε, ε, ήρθε, ήταν η ώρα της διαπραγμάτευσης είχε ενεργειακού πόρους. Ήταν ένα άρθρο το οποίο έτυχε ιδιαίτερης προσοχής όταν ε, στην Βουλή των Λόρδων δώσαμε προσοχή και εξετάσαμε αυτό το θέμα. Περιπλέκει όμως το θέμα καθότι ακούσαμε προηγούμενα. Έχω τρεις ερωτήσεις λοιπόν σχετικά με αυτά. Πρώτα απ' όλα, δίνοντας συνέχεια στο σημείο το οποίο αναφέρθηκε από πλευρά του εισηγητή κυρίου Σάριους Βόλσκι για τις συζητήσεις ε, που διεξάγονται αυτή τη στιγμή μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την ενεργειακή ασφάλεια από ό,τι γνωρίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να συμπεριληφθεί στον κανονισμό μια δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονηθεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις ε, ενεργειακές μας ανάγκες. Τι συμβαίνει τώρα. Εδώ θα έπρεπε από πλευρά ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πιστούν τα εθνικά κοινοβούλια να ασκήσουν πίεση στα, ε, στις κυβερνήσεις ώστε να παραμείνει αυτό μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του τριμερού στον διαλόγου δεύτερη ερώτησή μου αφορά την οδηγία για τις, ε, τα ε, πετρελαϊκά αποθέματα. Ζητείτε, απαιτείτε από τα κράτη-μέλη μέχρι το 2012, ε, τα τέλη του 2012, να έχουν υψηλότερα πετρελαϊκά αποθέματα. Διερωτώ με, ποια είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά αυτά τα αποθέματα. Και εν τέλει θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση μεταξύ όσον αφορά την αμφίδρομη δράση, την επιρροή των θεμάτων της ενεργειακής, του ενεργειακού ανεφοδιασμού και της αηφορίας, της βιωσιμότητας. Μακροπρόθεσμα η ε, μείωση των ε, πηγών άνθρακα θα πρέπει να μειώσει την εξάρτησή μας από εξωτερικές πηγές ενέργειας. Υπάρχει όμως κίνδυνος ε, βραχυπρόθεσμα η επικέντρωση σε θέματα ασφάλειας να μειώσει τις προοπτικές μας να επιτύχουμε Έχουμε την βιωσιμότητα. Η διασύνδεση μεταξύ αυτών των δύο θεμάτων είναι αρκετά σημαντική και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σα uh, Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Καθώς είμαι μέρος της διαπραγματευτικής ομάδας με το Συμβούλιο για την Ασφάλεια Ανεφοδιασμού Φυσικού Αερίου, πιστεύω πως αυτό δεν είναι το βασικό εμπόδιο εδώ. Υπάρχουν κάποια ζητήματα, υπάρχουν ε, μικρότερα προβλήματα που εν γέννη αφορούν το ρόλο της Κομισιόν και τη δυνατότητά της να εφαρμόσει και ίσως να σχεδιάσει εκ από τα εθνικά προγράμματα για τον ανεφοδιασμό σε φυσικό αέριο. Θα τα συζητήσουμε μέσα στι επόμενε δύο-τρει εβδομάδε. Αυτά είναι πρώτε μου απαντήσει. Ο κύριο Ένση από το ε, Ρωμανικό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ. Το θέμα της ασφάλειας ε, τη ανεφοδιασμού σε ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί κάτι τέτοιο, γιατί αν καταναλώνουμε λιγότερο θα έχουμε περισσότερη ενέργεια στη διάθεσή μας. Η ευρωπαϊκή διάσταση μπορεί να το καταφέρει αυτό. Έχουμε κανονισμούς, έχουμε αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Η εφαρμογή είναι πολύ σημαντική, σημαντική για να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα σε ενέργεια. Έχω ίσως κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να μας προβληματίσει το κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να πιστούν για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τους προσφέρει ενεργειακή ασφάλεια Νομίζω πως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να πιστούν δηλαδή τα ίδια τα κράτη-μέλη. Ίσως κάθε κρατός μέλος να πρέπει να συμβάλλει σε αυτή την εσωτερική αγορά ενέργειας και κάθε χώρα να εξειδικευτεί σε ένα είδος ενέργειας. Η ύπαρξη των μιας μελλοντικής κοινότητας ενέργειας ε, προϋποθέτει τη λήψη υπόψη των ε, γεωγραφικών, κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών, ώστε κάθε περιφέρεια να μπορεί να προσφέρει κάτι στην αγορά ενέργειας. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι για το γεγονό ότι δημιουργώντα μια κοινή αγορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να εξασφαλίσει την ενεργειακή ε, τον ανεφοδιασμό σε ενέργεια για κάθε χώρα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες κάθε χώρας, να βρούμε λύσεις που θα εφαρμόσουμε όταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργεια θα γίνει μια πραγματικότητα. Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο στεναρή ενεργειακή πολιτική. Μια Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την Ενέργεια δεν δικαιολογείται παρά μόνο από το πνεύμα της αλληλεγγύης και μόνο αν συμπεριλαμβάνει όλα τα κρατημέλη, όποια και είναι η κατάστασή τους και η δυνατότητά τους να συμβάλλουν σε αυτή την εσωτερική αγορά. Η προσπάθειά μας θα πρέπει να είναι συλλογική και δεν μπορεί να αφορά μόνο μια ομάδα χωρών, ακόμα και αν αυτές οι χώρες αποτελούν τον οικονομικό πυρήνα της Ένωσης. Θα έπρεπε να είναι προσπάθεια όλων των χωρών μελών, των 27 χωρών μελών, διότι κάτι τέτοιο αντιπροσωπεύει έναν τρόπο Συγκεκριμένοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή επιτυχία μας εξαρτάται από τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. κύριος Λικηγέ από την Γαλλική Εθνοβουλή. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον φίλο μου Ζάιρο Σβόρσκι για την εισαγωγή του και να του πω ότι συμφωνώ πλήρως. Θα ήθελα να επιμείνω στο γεγονός ότι εδώ ομιλούμε για ένα πολύ βασικό πρόβλημα για την Ευρώπη διότι πρόκειται για την ανεξαρτησία της και όλοι εμπλεκόμαστε και ενδιαφερόμαστε για αυτό το θέμα και ιδιαίτερως οι χώρες ε, οι ανατολικές και της κεντρικής Ευρώπης και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στην έκθεση η οποία μας έχει δοθεί μαζί με το φάκελο βλέπουμε ότι η ανεξαρτησία μας διακυδεύεται όσον αφορά τη Ρωσία. Και στο θέμα αυτό όπως και σε πολλά άλλα γίνονται πολλές εκθέσεις, νομίζω ότι κάνουμε ε, ε, πρόοδους, δεν είμαι όμως βέβαιος. Και τέλος πιστεύω ότι διέφτασε η ώρα να ασχοληθούμε με συγκεκριμένα θέματα και να ξεπεράσουμε και να βελτιώσουμε την αξιολόγηση των προβλημάτων τα οποία είναι εθνικά και μας διακρίνουν τους μεν από τους δε. Στη στρατηγική αυτή την οποία εξετάζουμε ε, σε σχέση με τη Ρωσία αλλά και σε σχέση με τις ενεργειακές παραγωγές μας διότι ξέρω ότι το θέμα αυτό είναι ταμπού διότι ε, σε άλλες χώρες συζητείται αλλού λιγότερο το θέμα αυτό το ταμπού είναι το πυρηνικό και για να μπορέσει η Ευρώπη να επιτύχει πρέπει να αποδεχθεί στο σύνολό της την πυρηνική ενέργεια. Ξέρω ότι υπάρχουν ντροπέ ταμπού, αλλά όταν έχουμε πρόβλημα ανεξαρτησίας ενεργειακής πρέπει να διασφαλίσουμε στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών ε, και αυτών που σήμερα δεν θέλουν και αντιδρούν, διότι αυτή είναι μία ανάγκη ε, ανεξαρτησίας. Και θέλω να κάνω και μία τρίτη παρατήρηση. Προηγουμένως ήταν ενδιαφέρον Πρόκειτο για δύο νομικούς οι οποίοι ε, είχαν στραφεί περισσότερο προς αυτήν τη σκοπιά. Αλλά τώρα δεν είναι θέμα να συζητάμε νέες συνθήκες και νέα κείμενα. Το ερώτημα είναι αν έχουμε την πολιτική θέληση της αυτονομίας ε, από ενεργητικής σκοπιάς. Διότι έχουμε το άρθρο 194, έχουμε τη δυνατότητα της ενισχυμένης συνεργασίας και πιστεύω ότι πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Και πρέπει να σας πω ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε η πρώτη προσπάθεια ενισχυμένης συνεργασίας σε ε, δικαστικά θέματα και πιστεύω ότι είναι καλό διότι ε, επέτρεψε σε 14 κράτη που ε, συνένεσαν την Παρασκευή στα θέματα διαζυγίου στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας να προχωρήσουν διότι όχι δεν θα προχωρήσουν σε διάφορα θέματα αλλά θα μπορέσουν να προωθήσουν διάφορα από αυτά και να προσκαλέσουν και τα υπόλοιπα κράτη να ακολουθήσουν την πορεία αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι από πλευρά κειμένων έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τώρα μία πεπισμένη πολιτική θέληση για ένα τόσο βασικό θέμα για την Ευρώπη, εξίσου σημαντικό όσο και την Ευρώπη της κρίσεως και της, ε, της ασφαλείας και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να το προωθήσουμε όχι με νέα κείμενα αλλά με δεδηλωμένη θέληση συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Τόγια. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι να εκφράσω μια εκτίμηση για αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε συζητήσει ξανά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λίγο αντίθετα από τα όσα είπε ο συνάδελφος της, της, της Γαλλικής Βουλής πιστεύω πως ε, ένα τέτοιο είδος συνεργασίας ε, θα είναι ένα πρώτο βήμα για ενίσχυση με κάποιο τρόπο της, ε, του νομικού μας οπλοστασίου. Δεν ξέρω αν αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω μιας νέας συνθήκης, μιας ε, νέας συνθήκης ΕΚΑΧ ή με κάποιο άλλο τρόπο, γιατί πιστεύω τώρα ότι χρειάζεται ενίσχυση της νομικής βάσης. Δεν θέλω να υποτιμήσω την ε, πολιτική βούληση. Είναι πολύ σημαντική η λήψη μιας πολιτικής απόφασης και η ίδια η εμπειρία μου από αυτό το κοινοβούλιο λέει, όπως ε, εξελέγει πριν από πέντε χρόνια, είναι ότι όταν υπάρχει μια θέλουμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική ευρωπαϊκή, δεν υπήρχε η νομική βάση του 194 και ήταν μια τέτοια δυσκολία μετά από διάφορα γεγονότα, Ρωσία, Ουκρανία και άλλα επεισόδια, οδήγησαν έτσι ώστε στο εσωτερικό του Συμβουλίου να δοθεί εντολή στο... στην Κομισιόν για να τη πει να... που να λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει μια... να μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη ε, πολιτική. Δεύτερο πακέτο για την ενέργεια και για την εξασφάλιση των εφοδιασμών Ορισμένες Ορισμένε φορέ η πολιτική βούληση ξεπερνά την νομική, το νομικό εμπόδιο. Πιστεύω ωστόσο ότι σε αυτή τη φάση, επειδή χρειάζεται να προχωρήσουμε πιο γρήγορα σε επιλογέ περίπλοκε για αυτήν την κάθε χώρα, να έχουμε μια αξιολόγηση του νομικού πλαισίου θα ήταν απαραίτητο. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση και εύχομαι αυτή η πρωτοβουλία να κατευθυνθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ε, προς αυτή την πορεία. Δεύτερο σημείο που θέλω να θυμίσω αφορά ε, μία από τις τρεις λέξεις της ομάδας εργασίας μας. Διαφοροποίηση. Πολύ συχνά όταν μιλάμε για ασφάλεια σκεφτόμαστε περισσότερο να εξασφαλίσουμε τους ελεύθερους οδούς προς τις ε, προμήθειε, ε, του διαδρόμου, την αλληλεγγύη κτλ. Αλλά πιστεύουμε και σκεφτόμαστε τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Όμως για την ασφάλεια και την ε, μη εξάρτηση ή μάλλον τη μεγαλύτερη αυτονομία σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση εξάρτησης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη από ορισμένε χώρε, όχι μόνο τη Ρωσία, αλλά και άλλε χώρε ασιατικέ ή αφρικανικέ, είναι ακριβώ να στοχεύσουμε στην διαφοροποίηση. Μπορεί να είναι κάτι το μπανάλ να ακούγεται, γιατί όχι μόνο το, στο Κοινοβούλιο αλλά και με την Κομισιόν αποφασίσαμε το πακέτο το 2020-2020 αλλά και γιατί θα πρέπει πιο συχνά να, μάλλον, να μην υποτιμούμε την, ε, το εύρος αυτής της απόφασης. Πολύ συχνά ε, χαρακτηρίζονται ως ε, ουτοπικές οι ευρωπαϊκές επιλογές. Όχι, δεν είναι κάτι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θέλουμε να στοχεύσουμε στη διαφοροποίηση και κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις οποίες οι στόχοι που προβλέπονται ακόμα και για τη δική μου χώρα, δηλαδή να τους φτάσουμε μέχρι το 2020, είναι περίπλοκοι στόχοι. Ελπίζω και εύχομαι, όπως το κάνουμε τώρα με ορισμένε οδηγίες σε σχέση με την ενεργειακή επάρκεια που αποθύμησε και ο συνάδελφος και την ενεργειακή εξοικονόμηση, ότι θα πρέπει να υπάρξουν διάφορες στάδια

δεσμευτικά ενδιάμεσα. Γιατί αν δεν υπάρξουν τέτοια στάδια, δεν θα ε, καταφέρουμε να πετύχουμε του στόχου του 2020. Να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, λέγοντα ότι όταν μιλάω για διαφοροποίηση, δεν σκέφτομαι απαραίτητο ε, την απέτηση τη εξάπλωση τη πυρηνική ενέργεια ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλε τι χώρε. Είναι μια επιλογή εθνική. Γιατί διαφοροποίηση συζητείται σε όλε τι χώρε και στη χώρα μου η πλειοψηφία ακολούθησε μια πορεία. Δεν συμφωνούν όλοι οι το πολιτικό φάσμα. Εγώ δεν συμμερίζομαι εις βάθος αυτή την ε, επιλογή, αλλά πιστεύω ωστόσο πως μια μεγάλη διαφοροποίηση, μεγάλη δέσμευση για αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα για να έχουμε εξοικονόμηση, καθώς και η χρήση όλων των τεχνολογικών ε, ε, δυνατοτήτων που προσφέρονται σήμερα, μας επιτρέψουν να έχουμε ένα τέτοιο μείγμα διαφοροποίησης, ώστε να έχουμε ασφάλεια στον ανεφοδιασμό, να μην εξαρτώμεθα χωρίς να αποκλείουμε και την πυρηνική ενέργεια στο πλαίσιο αυτών των επιλογών να υπογραμμίσουμε την εξωτερική πολιτική. Εδώ έχουμε ξεκινήσει μια θεσμική μεταρρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που σήμερα βλέπουμε να έχουμε μια προσωπικότητα του, όπως αυτού του Ευρωπαίου ε, Υπουργού Εξωτερικών. Πιστεύω πως θα πρέπει να συνδέσουμε τις ενέργειες σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης με αυτή την πτυχή της ε, ενεργειακής ασφάλειας που συμπεριλαμβάνει και αυτή την πτυχή σε εμπορικό επίπεδο αλλά και σε στενότερες σχέσεις με όλες αυτές τις χώρες. Σας ευχαριστώ. Επόμενο είναι ο κ. Κόζιτς από την Κροατία. Σας ευχαριστώ. Θα έλεγα ότι η ασφάλεια η ενεργειακή μπορεί επισήμως να οριστεί ως ένα είδος γεωπολιτικού παιχνιδιού σημαίνει ότι ο χαρακτήρας του προβλήματος είναι πολύ περισσότερο παιχνίδι παρά μια απλή και ξεκάθαρη πολιτική. Αν δεχτούμε ότι κάτι τέτοιο ε, ισχύει, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο χαρακτήρας αυτού του παιχνιδιού είναι μηδενικός. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια κατάσταση win-win, όπου όλοι κερδίζουν. Αλλά όταν αγωνιζόμαστε για κοινού διαδρόμου ή κοινέ πηγέ φυσικού αερίου ή πετρελαίου, ανταγωνιζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο. Κεντρική Ασία, καλύτερο δείγμα. Τουρκμενιστάν, νέε πηγέ, Κίνα, Ινδία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, τσακώνονται για την επιρροή τους και για τον αντίκτυπό τους και για το ποιος θα μπορέσει πρώτος να πάρει αυτούς τους πόρους στον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι έχουμε πραγματικούς περιορισμούς, περιορισμούς στον καθορισμό κοινή ενεργειακής πολιτικής, διότι μέσα σε αυτό το παιχνίδι έχουμε συγκρούμενα συμφέροντα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρουμε να ελοχιστοποιήσουμε τις συγκρούσεις αυτές, τις αντιπαραθέσεις και να δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε κοινούς στόχους ε, ή όταν μιλάμε για την τεχνολογία. Ο τσακωμός αφορά διάφορες εταιρείε. Ποιος δηλαδή θα ηγηθεί, ποιος θα καταφέρει να βρίσκεται στην αιχμή στο επίπεδο τεχνολογίας. Γιατί μια εταιρεία αν είναι η ε, ηγετική, προηγείται, θα έχει στρατηγικό πλεονέκτημα στην αγορά. Το κεντρικό πρόβλημα λοιπόν είναι να καταλάβουμε τι είδους παιχνίδι παίζεται. Διάφορε υπηρεσίε αντικατασκοπία ενεργούν στον τομέα τη ασφάλεια ανεποδιασμού ενέργεια και αυτό ο ορισμός μιας συνολικής προσέγγισης θα πρέπει να γίνει για να δούμε τι είδους περιορισμούς έχουμε να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά τον καθορισμό μιας κοινή ενεργειακής πολιτικής. Και δίνω το λόγο στη Συμπρόεδρο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάμπους από τη Σλοβενία είναι επόμενος θα μιλήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που δώσατε τον λόγο. Αξιότιμοι συνάδελφοι, επαΐοντες, με μεγάλη χαρά παρακολουθήσαμε τη συζήτηση. Είναι εξαιρετική η συζήτηση και τα θέματα. Και πρέπει να πω ότι την κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υποστηρίζω. Είναι όμως σημαντικό οι συνάδελφοι το ότι έθεσαν, ε, ε, έθιξαν ένα θέμα ιδιαίτερη σημασίας. Ιδιαίτερα αυτό δηλαδή των επενδύσεων στα ενεργειακά θέματα από πλευρά των κρατών μελών μας. Εδώ θα πρέπει με ιδιαίτερη σύνεση να δράσουμε γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα επιμέρους κράτη-μέλη έχουν διαφορετική ανάπτυξη και παρόλα αυτά πρέπει να βρούμε ένα κοινό παρονομαστή για αυτές τις πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να πω ότι είναι αναγκαίο να εκπονήσουμε παραμέτρους και συντελεστές που θα διευκολύνουν την αναζήτηση αυτού του κοινού παρονομαστή, ώστε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να είμαστε σωστοί στις δράσεις μας και με ίσα δικαιώματα και ίση δυνατότητα πρόσβασης να μπορούν τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτά τα βήματα προς την κοινή ενεργειακή πολιτική με τον ίδιο στόχο και κοινή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ. Ο Έντμον Βίτπρετ είναι επόμενος από τη Γερουσία της Πολωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ το Γιάτσεκ Σάρους Βόλσκι για την έξοχη εισαγωγή που έκανε και για τη συζήτηση που διεξάγεται. Ακούγοντας τη συζήτηση αισθάνομαι ότι όλοι σε κάποιο βαθμό έχουν δίκιο. Αλλά είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς μπορούν να συμφιλειωθούν όλες αυτές οι αποκλίνουσες απόψεις. Ένα πράγμα είναι βέβαιο. Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα ή η κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική είναι ζωτική σημασία και θα πρέπει να βασίζεται σε αλληλεγγύη. Η Πολωνία ήταν από τι πρώτε χώρε που υποστήριξε ένα κοινό σύστημα ενεργειακού εφοδιασμού. Και αυτό λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων που επικρατούν στην Πολωνία, πολιτικών συνθήκων και περιορισμένων πόρων όσον αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η ιστορική μας εμπειρία είναι τέτοια που ε, μας κάνει να διστανόμαστε ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, ενδεχόμενοι κίνδυνοι και θεωρούμε ότι μια κοινή πολιτική παρέχει κάποιες δυνατότητες. Βλέποντας τον τίτλο της ομάδας εργασίας «Ενεργειακή ασφάλεια, ποικιλομορφία, αλληλεγγύη και αλληλεξάρτηση όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό» δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε για αυτά τα τρία στοιχεία και να τα θεωρούμε ότι ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Διότι και τα τρία στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν τμήμα της εξίσωσης δεν έχει νόημα να έχει κανείς ποικιλομορφία πηγών αν δεν υπάρχουν δίκτυα ε, μετάδοσης της ενέργειας. Να πηγαίνει η ενέργεια εκεί που χρειάζεται. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για αλληλεγγύη αν δεν βελτιωθούν οι υποδομές και αν δεν αναπτυχθούν χώροι αποθήκευσης για την ενέργεια που παράγεται και εισάγεται. Πρέπει να είναι κανείς σίγουρος ότι ο εφοδιασμός ενέργεια και αποθήκευση ε, είναι ασφαλή από πολιτικά παιχνίδια. Ποικιλομορφία, αλληλεγγύη και αλληλεξάρτηση και τα τρία στοιχεία είναι ζωτική σημασία όσον αφορά την ποικιλομορφία. Θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι κομμάτι της εξίσωσης Αναφερθήκαμε στην εξοικονόμηση ενέργειας, αποδοτική χρήση ενέργειας, εκπαιδεύσεως του κόσμου, έρευνα για εξοικονόμηση σε ενέργεια και κάποιες αποφάσεις ελήφθησαν στην Πολωνία μάλιστα ελήφθησαν αποφάσεις υπέρ της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και θα λειτουργεί μια μονάδα πυρηνική μέχρι το 2020. Το ερώτημα είναι μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτόν και αυτό είναι το πρώτο ερώτημα προς τον Γιάτσεκ Ζαρουζόλσκι. Γιάτσεκ Σαρουσβόλσκι, συγγνώμη. Ποιο είναι το πολιτικό μας όραμα. Ο κύριος Σαρουσβόλσκι αναφέρθηκε στο όραμα και στην πολιτική βούληση πρέπει να υπάρχει αλλά νομίζω ότι ακόμα ψάχνουμε το όραμα. Πολύ μάλλον δεν την πολιτική βούληση. Ακόμα και όταν υπάρχει όραμα, καμιά φορά λείπει η πολιτική βούληση για να εφαρμοστούν οι κανόνες που έχει θεσπίσει. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Συμφωνώ με εκείνους που διαρωτώνται για το πώς θα μπορέσουμε να συμφιλιώσουμε τις διάφορες αντιφάσεις που υπάρχουν. Οι μελέτες έχουν καταδείξει ότι τα διάφορα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά συμφέροντα και είναι δύσκολο να βρεθεί κοινός, ελάχιστος κοινό παρονομαστής ούτως ώστε να συμφωνήσουν οι χώρες. Και εντός κρατών μελών υπάρχουν επιχειρήσεις και επιχειρήσεις καμιά φορά έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Όταν λοιπόν αναφερόμαστε στην αλληλεγγύη και είναι το ερώτημά προς το Γιάτσεκ Ποιο θα πληρώσει για αυτή την αλληλεγγύη, αυτό το ερώτημα. ποιο πληρώνει. Ευχαριστώ κύριε Βίτπρατ. Η κυρία Ζαν Μπισέτ της ε, Γαλλικής Γερουσία είναι η επόμενη. Ο κύριος. Ε, λυπούμε, λέει η Πρόεδρος, ο κύριος λοιπόν. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα το ενεργειακό στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από ε, εξαιρετική περιπλοκότητα. Όλοι οι στόχοι, ό,τι συνδέονται ε, στενά μεταξύ του. Είναι πολύ ευαίσθητο να ασκηθεί μια πολιτική στο δεδομένο τομέα, χωρί να λαμβάνουμε υπόψη όλο το θέμα συνολικά, το ενεργειακό. Για να πάρουμε παράδειγμα το θέμα μα, την ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό, εξαρτάται άμεσα από τι ενδογενεί ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και από την έρευνα για καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα επίσης εξαρτάται από τη δημιουργία ενίας αγοράς ενέργειας που βασίζεται σε ένα δίκτυο ευρωπαϊκό μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου. Όμως οι λύσεις δεν είναι προφανείς. Έτσι, η ανάπτυξη των νεωσίμων πηγών λύσει δεν είναι κάτι συνώνυμα απαραίτητα με μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αναπτυξη των νεοσυμων πηγων ενεργειας δεν ειναι κατι συνωνυμα ενέργεια η, η νέα γενιά μπαταριών χρησιμοποιούν σπάνια μέταλλα σπάνια, σπάνια ορυκτά που κυρίως τα εξάγει η Κίνα. Άρα δεν υπάρχει αυτόματο συσχετισμό μεταξύ ανανεωσίμων πηγών ενεργεία και ενεργειακού ασφαλού εφοδιασμού. Ακόμα και αν η ενέργεια αποτελεί ένα, ε, αυτά τα είδη ενεργειών αποτελούν σημαντικό τμήμα τη λύση. Θα επανέλθω τώρα στο θέμα τη αλληλεγγύη που αναφέρθηκε. Βεβαίω όλοι συμφωνούμε. Θα πρέπει να ισχύσει η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, κυρίως σε περίπτωση κρίσεως όσον αφορά τον εφοδιασμό ενός κράτους μέλους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί από άκρως ολοκληρωμένα δίκτυα που επιτρέπουν τη μετάφορα ηλεκτρικής ενέργειας ή καυσίμων ε, μέσω της Ευρώπης. Αυτά τα δίκτυα επίσης καθίστανται αναγκαία στο βαθμό που το τμήμα των ανανοσίμων πηγών ενέργειας αυξάνεται, η ολική ενέργεια δεν έχει σταθερή παραγωγή και προβλέψιμη παραγωγή για ηλεκτρική ενέργεια, θα πρέπει να αντισταθμίζεται από μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας αν υπάρχει μείωση παραγωγής από την αιωλική. Αλλά θα πρέπει αυτή η αρχή της αλληλεγγύης να μην επιτρέπει σε μια χώρα να χαλαρώσει τις επενδυτικές της προσπάθειες βασιζόμενη στην παραγωγή των γειτόνων σε περίπτωση ανάγκης. Αυτό που υπενόησε η πρόσφατη παρέμβαση του συναδέλφου όσον αφορά το θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Η πρόταση κανονισμού για τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο που εξετάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να φροντίσει γι' αυτό. Τώρα που μιλάμε πολύ για οικονομική διακυβέρνηση, η ενεργειακή διακυβέρνηση θα πρέπει να συζητηθεί, είναι θεμελιώδου σημασίας Αντίθετα, η σύγκληση των πακέτων των ενεργειακών των ευρωπαϊκών δεν θα πρέπει να είναι ένα στόχο το να πετύχουμε πάση θυσία. Συναρτήση τη γεωγραφία, των ωφελημάτων, θα πρέπει κάθε κράτο μέσο καθορίσει το δικό του πακέτο το ενεργειακό. Και αυτή η ποικιλομορφία, κάθε χώρα θα προωθεί μια συγκεκριμένη πηγή ενέργεια. Λοιπόν, αυτή η ποικιλομορφία μπορεί να ευνοήσει τη δημιουργία μια κοινοτική ε, ενεργειακή κοινότητα. Ας πούμε μπορεί να είναι μια χώρα που θα προωθεί την ολική ενέργεια και μπορεί να χρειάζεται ε, ηλεκτρική ενέργεια από κάποια χώρα που παράγει μέσω άνθρακα, φυσικού αερίου ή άλλων πηγών ενεργειών. Ε, έτσι μπορεί να επιτευχθεί η κοινότητα, η ενεργειακή. Σε χρόνια θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή και νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσει η προσπάθεια ήδη, χωρίς να χάνουμε χρόνο. Χρειάζεται ενισχυμένη συνεργασία εκτός των συνθήκων Νομίζω ότι είναι η σημερινή λύση, η πιο καλή λύση σήμερα, υπό τις ε, παρούσες συγκυρίες. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος ε, ο μιλητής είναι ο κύριος Σαφίφ Ντεμακίδαν από την Τουρκία. Ευχαριστώ. Ε, κύριοι Πρόεδροι, Συμπρόεδροι, ε, χαίρομαι που είμαι εδώ και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ισπανικό Κοινοβούλιο για την ε, ε, πρόσκλησή τους. Είμαι πρόεδρος της ε, τουρκο-ισπανικής ε, οργάνωσης ε, βουλευτών και φιλίας και γι' αυτό προσεκλήθη. Όταν μιλάμε όμως για ασφάλεια ενέργειας δεν μιλάμε μόνο για την Ευρώπη την οποία πρέπει να σκεφτόμαστε αλλά όλο το κόσμο, όλη την Ιφίλιο όσον αφορά την ασφάλεια όπως άλλωστε αναφέρετε στην έκθεσή σας διότι όταν θα φτάσουμε το 2030 θα υπάρχει 40% αύξηση της ε, ε, ενεργειακής ζητήσεως σε σχέση με σήμερα και η Τουρκία παραδείγματος χάρη σε 15 χρόνια θα διπλασιάσει την κατανάλωσή της. Άρα οι χώρες της Ευρώπης και η ασφάλεια παροχή τους και η ασφάλεια παροχής ε, ενεργείας της Τουρκίας πρέπει να αξιολογηθούν από κοινού. Σαν υποψήφια χώρα Έχουμε κληθεί σε αυτή την συνεδρίαση και θα ήθελα εδώ να παρουσιάσω ένα από τα παράπονά μου και ε, να πω ότι ε, παρόλο που η ενέργεια και η ρύθμιση ενεργειακή της Τουρκίας συνάδει πλήρως με το ενεργειακό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ατυχώς δεν ε, υπάρχει δεν υπάρχουν μέτρα και στα κοινά και δεν έχει ανοίξει το κεφάλαιο της ενεργείας που θα έπρεπε να το ανοίξουμε σε λεπτομερείς συνεδριάσεις διότι όταν μιλάμε για ασφάλεια της ευρωπαϊκής ενέργειας δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την Τουρκία που είναι σε κάποιο χώρο όπου 72% όπου βρίσκονται, ε, που βρίσκεται κοντά σε 72% των ε, ενεργειακών αποθεμάτων ε, από πλευράς πετρελαίου και αερίου, δηλαδή την κεντρική Ασία. Για να υπάρχει λοιπόν η ποικιλομορφία της παροχής ενεργείας στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε και την Τουρκία πλέον της ε, Αλγερίας και της Ρωσίας. Χρειαζόμαστε τους αγωγούς που διέρχονται και ορισμένοι από αυτούς έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάποιος συνάδελφος ανεφέρθη στον Ναμπούκο που έχει ήδη υπογραφεί η διακυβερνητική συμφωνία. Λέγεται ότι το Ναμπούκο δεν θα έχει, ο ε, αγωγός Ναμπούκο δεν θα έχει επαρκή παροχή αερίου όταν θα φτάσουμε το 2018 θα υπάρχει πολύ μεγάλη παροχή και πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε ε, ίσως όχι να καλύψουμε τις ανάγκες της Ευρώπης διότι έως τότε ε, θα υπάρξει μία αύξηση της ζητήσεως αερίας 100 μέχρι 200 δισεκατομμύρια κυβικά αλλά ε, το Ναμπούκο είναι μία από τις, ε, τους αγωγούς, ένας από τους αγωγούς που θα χρησιμοποιηθούν και η ε, Τουρκία, η Ελλάδα, η Ιταλία συνδέονται δηλαδή εμείς ήδη προωθούμε το αέριο προς την Ελλάδα και από εκεί μπορεί να πάει στην Ιταλία και στις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να, να ληφθεί υπόψη συλλογικά ότι η Τουρκία πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα πλήρες μέρος και να ανοίξουμε το κεφάλαιο της ενεργείας προς διαπραγμάτευση. Και τελειώνω. Μια άλλη πληροφορία όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια είναι η διασύνδεση ηλεκτρισμού μεταξύ Τουρκίας και της Ευρώπης που έχει ήδη γίνει και ήδη εφέτος θα λειτουργήσει το σύστημα που θα επιτρέπει να υπάρχει ανταλλαγή ηλεκτρισμού μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας. Ανανεώσιμες πηγές ενεργείας που ε, ελέγχθη για το 2020 μιλήσαμε για 20% αύξηση αποδοτικότητας και μείωση κατά 20% των ε, εκπομπών ε, αερίων αλλά εμείς ήδη σύντομα θα έχουμε προχωρήσει και θα μπορεί η Ευρώπη να αγοράζει περισσότερη πράσινη ενέργεια από την Τουρκία όταν θα έχουν συνδεθεί. Ε, είμαστε ενάντια στην πυρηνική ενέργεια αλλά πιστεύω ότι θα είναι μία από τις ενεργειακές ε, πηγές στην Ευρώπη και παντού και είναι ένα θέμα που αρχίζει να συζητείται για ε, την οικοδόμηση ε, των ε, πρώτων πυρηνικών σταθμών που θα λειτουργήσουν μέσα στα επόμενα 12 χρόνια. Ευχαριστώ τον κύριο Ντεμερκύραν. Ε, παρακολουθούμε την εξέλιξη της Τουρκίας και ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος, ένας εκπρόσωπος της Σλοβακίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε η δημοκρατία της Σλοβακίας είναι ένα κράτος που τα μέγιστα από την κρίση του φυσικού αερίου επλήγει. Είχαμε φτάσει στα όρια του blackout και γι' αυτό όλα τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας του ανεφοδιασμού μας με ενεργειακά προϊόντα έχει τεράστια σημασία. Θέλω να τονίσω ότι ήταν η αλληλεγγύη που μας βοήθησε να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας ε, και από την Γερμανία και ε, οι προσπάθειες ε, που ανελήφθησαν έδωσαν τη δυνατότητα να λυθούν τα προβλήματα παροχής φυσικού αερίου. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα δεν θα μπορούσαμε να είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Αυτά όλα ήταν πάρα πολύ αισθητά στην οικονομία και πρέπει μέχρι σήμερα ακόμα να αγωνιζόμαστε με τις επιπτώσεις της προηγούμενης κατάστασης. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα θέματα των διμερών παροχών, της διμερούς παροχής ενέργειας. Θέλω να πω ότι παραμένει και υφίσταται μείζον πρόβλημα αυτό. Παραμένω στο φυσικό αέριο. North Stream, South Stream, Nabucco λοιπά Υπάρχουν διάφορες ε, φυσικά δυνατότητες και υπάρχουν και διαπραγματεύσεις από πλευράς ε, των κυβερνήσεων. Έχουμε και ε, ιδιωτικές εταιρείες και τίθεται το ερώτημα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση δυνατότητα να συμμετάσχει καν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις για την παροχή συγκεκριμένου όγκου ενεργειακών προϊόντων. Εδώ θέλουμε να, θέλω να αναφέρω ότι το δυναμικό για παράδειγμα της, ε, του αγωγού της ε, Ουκρανίας 100 εκατομμύρια κυβικά ε, μέτρα έχει μειωθεί και αυτό το δυναμικό μόνο σε, κατά 90% το εκμεταλλευόμαστε και αυτό αν συρρυκνωθεί θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δική μας οικονομία. Ο ενεργειακός ανεφοδιασμός και η ασφάλειά του δεν είναι μόνο τα θέματα τα οποία αφορούν αυτή την πτυχή. Είναι ένα ευρύτερο θέμα το οποίο συνδέεται με την κατανάλωση ενέργειας. Είναι και ένα θέμα της παροχής ηλεκτρικής, ε, ηλεκτρικού ρεύματος. Κάνουμε λόγο και για μελλοντικές ε, εξοικονομήσεις 20% στο ύψος του 20%, 20-20-20. Έχουμε περιορισμένα κονδύλια, περιορισμένες δυνατότητες και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει στο μέλλον να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ε, πυρηνική ενέργεια, στην ατομική ενέργεια ως δυνατότητα ε, παραγωγής ε, ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι η μόνη εφικτή λύση η οποία μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στην, στην αυξανόμενη ζήτηση. Ο συνάδελφος από την Τουρκία έθιξε το θέμα της ασφάλειας Αναφέρθηκε το θέμα της ασφάλειας, όμως η πυρηνική ενέργεια είναι η φθηνότερη πηγή ενέργειας. Πρέπει ιδιαίτερη προσοχή να δώσουμε στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας για να είμαστε επιτυχείς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν τι συμβαίνει. Υπάρχουν αρκετά μεγάλες διαφορές μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών. Στην ε, δημοκρατία μας, στη Σλοβακία, είχαμε ακόμα και κιόλας πριν από δύο χρόνια μια κατά 40% μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, απόδοση σε σχέση με τα κτίρια μας και την πολιτική μας έναντι των ε, ανεπτυγμένων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται το θέμα και της συνεργασίας εδώ συνεργασίας. Θα πρέπει να έχουμε τις πιο καλές προτάσεις και προσεγγίσεις για το μέλλον. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής είναι τώρα ο κ. Άνσετ. από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θέλει κάποιος ακόμα να μιλήσει, ναι, παρακαλώ, μπορείτε να γράψετε τα ονόματά σας. Ο κύριος Γκρίτερ από το Ευρωκοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Γιάννη Σάιρους Βόλτ διότι τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για το θέμα της ασφάλειας των ενέργεια εδώ και αρκετά χρόνια. Το 2007 σχετική έκθεση αποτέλεσε το βασικό συστατικό που έπεισε την κοινότητα να συμπεριλάβει τη διάταξη περί ενέργειας στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Όλοι γνωρίζουμε ότι το θέμα της ενέργειας έχει να κάνει με τη γεωπολιτική και όλοι οι μεγάλοι παίκτες προσπαθούν να καπαρώσουν ένα κομμάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παρακολουθεί παθητικά. Πρέπει να εξασφαλίσει την ε, απαραίτητη ενέργεια και το κατάλληλο μείγμα ενέργειας ώστε να μπορούμε να έχουμε όλοι μια μεμονωμένη ξεχωριστή προσέγγιση. Το ερώτημά μου στον κύριο Βόλσκι είναι τι ρόλο έχουν να παίξουν οι γείτονές μας στην ασφάλεια ανεφοδιασμού ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλώ για τους ανατολικούς μας ε, γείτονες στην ε, ανατολική εταιρική σχέση τους εταίρους μας στην ε, πολιτική γειτνίασης γιατί για την ώρα ομφαλοσκοπούμε, δηλαδή κοιτάμε μόνο τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως έχουμε πολύ σημαντικούς εταίρους που έχουν μεγάλο ρόλο στην διανομή ενέργειας και είναι ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της σταθερότητας παροχής ενέργειας στην αγορά. Φυσικά και εστιάζουμε στους παραδοσιακούς πόρους ενέργειας, Μέση Ανατολή, Κασπία, Θάλασσα, Βόρεια Αφρική. αλλά βλέπουμε την ε, ανάδυση πιθανών νέων πηγών, νέων πόρων με πολύ σημαντικά αποθέματα. Και δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε σκεφτεί και την Αρκτική ως πιθανή πηγή ενέργειας για το μέλλον. Ποιος έχει τη δικαιοδοσία στην Αρκτική. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να επιληθεί πριν να μπορέσει κανείς να εκμεταλλευτεί τους πόρους. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα λοιπόν γιατί είναι θέμα που αφορά την Ορβηγία και τη Ρωσία. Ακούσαμε νωρίτερα σήμερα πως υπάρχει ένας βαθμός ε, κούρασης μετά από τη διεύρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έχει μειώσει την όρεξη για σύνταξη νέων συνθήκων. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή μας πώς θα ξεπεράσουμε αυτήν την κούραση, αυτήν την ε, απάθεια που μας έχει επηρεάσει και να κάνουμε κάτι στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής. Έχουμε βαρεθεί τη διεύρυνση, έχουμε βαρεθεί τους κανονισμούς. Οι δικοί μας έχουν τονίσει ότι ίσως χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία ώστε να λειτουργήσουν καλύτερα αυτές οι πολιτικές. Πάντως πιστεύω πως αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητή... είναι η κυρία Σιμώνα Βικάρη από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Εγώ Κοιτάξτε, θέλω να ακούσω ότι επακούσα αυτά που είπε ο Πρόεδρος, να έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση και ακολουθήθηκε. Οπότε οθήθηκα για να ζητήσω ξανά το λόγο για να πω κάποια σκέψεις που δεν έκανα στην πρώτη μου παρέμβαση. Ευχαριστώντας σας πολύ για αυτή την ημερίδα που μας προσφέρατε και την αυριανή. Και πριν και άλλες φορές να υπάρχει δυνατότητα να συναντηθεί. Έχουμε συναντηθεί και άλλες φορές, αλλά αυτή ήταν η πιο σημαντική συνάντηση. Και θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι τρόποι να συναντηθούμε και να προβούμε σε εμβαθύνσεις των θεμάτων. Όσον αφορά την Ιταλία, αφού ακούσαμε κάποια πράγματα, πρέπει να πω ότι η θέση επεκφράστηκε από τη Γαλλία και από την Πολωνία όσο με αφορά είναι απόψεις με τις οποίες μπορώ να συμφωνήσω. Δηλαδή ότι η φάση της συνεργασίας, όπως είπαν και οι νομικοί, είναι πιο χρήσιμη και πρακτική προσέγγιση αυτή τη φάση. Και η δεύτερη πρόταση, η ενιαία πράξη και η συνθήκη όπως το αποκαλέσουμε και αυτό χρήσιμο. Πρέπει να θεωρηθεί όμως σαν τελική φάση μιας διαδρομής. Κάτι στο οποίο καταφθάνομαι μετά από δουλειά, συνεργασία, πειραματισμό, αλληλεγγύη όσο την ασφάλεια. Ε, δηλαδή διαβουλεύσεις και όχι να ξεκινήσουμε προσπαθώντας να προλάβουμε κάτι. Θα πρέπει στην Ευρώπη επικρατεί αρχή ότι οι επιλογές θα πρέπει να ξεκινάνε από κάτω. Πράγματι, από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξεκινήσουν επιλογές. Το 2050, μέχρι το 2050, εν γέννη, θα έχουν θέσει όλα τα κράτη-μέλη σε στόχο να γίνει ο εφοδιασμός από φυσικές πηγές όπως σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και έχουμε 40 χρόνια μπροστά μας λοιπόν. Θα πρέπει να είναι φάση μετάβασης αυτή. Οι πηγές εφοδιασμού θα πρέπει να είναι επικοινωνόμορφες και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο βαθμό. Και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε με τις ε, πηγές που εξαντλούνται. Από αυτήν την οπτική γωνία, όχι επί την επιλογή της κυβερνήσεώς μου, αλλά του Ιταλικού λαού που υπερψήφισε το πρόγραμμα, το πυρηνικό πρόγραμμα που πρότεινε η κυβέρνηση, η πυρηνική ενέργεια, λέγω, είναι ενεργειακή πηγή η πιο σημαντική. Εδώ και μερικού μήνε και ο πρόεδρος τον είπα, ο Ομπάμα, παρουσίασε. Και την παραγωγή από πυρηνική ενέργεια, ενέργεια πυρηνική ενέργεια τέταρτης γενιάς, που θα πραγματοποιηθεί στην, στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ. Η Ιταλία ανήκει στου G8 αλλά σήμερα είναι η μόνη χώρα τον G8 που δεν παράγει ενέργεια από την πυρηνική ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για ελάχιστη αυτονομία μιας χώρας. Πρέπει να εξεταστεί σαν δεχόν πυρηνική ενέργεια. Είμαστε, είναι στα λίγα, έχουμε σε λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γαλλία πυρηνικό σταθμό και είναι παράλογο να μην έχουμε και στη μας χώρα. Ερώτηση προς συγκητή. Αναφέρθηκε στην οδηγία για το φυσικό αέριο. Ερώτηση. Αυτή είναι η νέα οδηγία για το φυσικό αέριο. Αν κατάλαβα σωστά. Προβλέπει υποδομές. Δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ κρατών μελών για να καταλάβουμε ποια προσπάθεια γίνεται σήμερα για να πετύχουμε ελάχιστο επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας. Σας ευχαριστώ, κυρία Βικάρη. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, ο κύριος Χάνες Σβόμποντα θα ήθελε να πει κάποιες, κάποια πράγματα πριν αποχωρήσει από τις Βρυξέλλες. Ο κύριος Σβόμποντα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύντομα σχόλια. Τρία, τον αριθμό. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Προείδρευσα αρκετών τέτοιων συζητήσεων. Είναι η πλέον ενδιαφέρουσα αυτή. Συμφωνώ με αυτά που μας είπε η κυρία Βικάρη. Τώρα, για την ε, ποικιλομορφία των πηγών ενέργειας. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να έχουμε πολλές πηγές ενέργειας. Αναφερθήκαμε, όταν μιλήσατε για τους πετρολαγωγούς, να μην ξεχάσετε ότι η καλύτερη διαφοροποίηση είναι η διαφοροποίηση των διαδρομών και των πηγών. Ο συνάδελφος από τη Σλοβακία νομίζω ότι αναφέρθηκε σε αυτό. Μπορεί η μία διαδρομή να αλλάξει να μειώσει την, τον εφοδιασμό μιας χώρας ή να μειώσει την ασφάλεια εφοδιασμού μιας χώρας αν αλλάξει τη διαδρομή. Δεν θέλουμε μόνο νέους, νέες διαδρομές αλλά και νέες πηγές. Δύσκολο μεν. Αλλά ο συνάδελφος από την Τουρκία είπε σαφώς ότι είναι σταδιακή διαδικασία. Αναφέρθηκε στον αγωγό Ναμπούκο για τη συνθήκη τώρα. Το έργο για μια συνθήκη που αλλάζει τη συνθήκη της Σαββόνας δεν θα ήταν κάτι πολύ επικοδομητικό. Από αυτά που υπόθηκαν, οι ομιλητές έχουν υπόψη τους συνθήκες που δεν είναι συνθήκες της Σαββόνας, αλλά τις συμπληρώνουν. Συμπληρωματική συνθήκη για αυτούς που είναι πρόθυμοι για κάτι τέτοιο. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε τις προσπάθειες του τελικού στόχου. Τελευταίο ερώτημα, δεν θέλω να αφαιρέσω τίποτα από αυτά που είπε και έκανε ο συγκητή σα διαπραγματεύσει για την εφοδιασμό σε φυσικό αέριο με το Συμβούλιο. Προσπαθούμε να ε, εφαρμόσουμε την εστροφή των ροών, τι διασυνδέσει, του αγωγού που είναι αναγκαίοι για να εξασφαλίσουμε το μέγιστο δυνατό εφοδιασμό σε φυσικό αέριο. Συγχώρηση που χρειάζεται να το κάνουν αυτό δεν είναι δυνατό αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κοινότητα πιστεύει ότι αυτού του είδου οι επενδύσει είναι σημαντικέ. Αυτό κάνουμε. Τι κάνουμε. Με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης αποφασίσαμε σε συναπόφαση με το Συμβούλιο και, την, και το Κοινοβούλιο να δοθούν αυτά τα κονδύλια. Δεν εκφανίζονται αυτά εκ το μηδενός, ήδη ακολουθείται αυτή η προσέγγιση. Πρέπει λοιπόν σε τρία χρόνια όλα τα κράτη-μέλη να εγγυηθούν ότι υπάρχει πλήρης εφοδιασμός φυσικού αερίου αν ένα από τα βασικά στοιχεία λείπει. Νι, μείον ένα είναι ο κανόνας. Και συμπεριλαμβάνεται. Χωρίς συγκεκριμένη ρητή αναφορά. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο της προσέγγισης για τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο. Δεν είναι κάτι θεωρητικό θα είναι νόμος που θα αποφασιστεί τον Ιούνιο. Αυτά τα τρία σχόλια έχω. Αυτά έχω συναγάγει από αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητώ συγγνώμη πρέπει να αποχωρήσω. Αλλά έχετε μια πολύ χαριτωμένη πρόεδρο και ο κ. Σαρσβόσκι, ο εισηγητής μας, θα δώσει τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κ. Σβόμποντα. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά δεν μπορώ ότι μπορώ να σας ανταγωνιστώ ούτε να ανταγωνιστώ τις δικές σας δεξιότητες. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Χερέρα. Ε, ε, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα πρέπει να πω με την περίληψη που έκανε ο κύριος και μόνο κάποια λίγα θέματα θα επισημάνω. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση που είναι τόσο ενδιαφέρουσα, αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, όταν έχετε η ώρα να καθορίσουμε τις θέσεις μας δεν πρέπει να ξεχάσουμε κάτι, μια αρχή πολύ σημαντική και αυτή είναι το ότι η Ευρώπη, στην Ευρώπη θέλουμε να αναπτύξουμε την ενεργειακή μας πολιτική παράλληλα με την περιβαλλοντική μας πολιτική. Γι' αυτό για να διασφαλίσουμε τον ενεργειακό ανεφοδιασμό δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο μία μόνο πηγή ενέργειας διότι μαζικά πηγές ενέργειας, ενέργειας υπάρχουν δύο αυτή τη στιγμή, τα ορυκτά καύσιμα και η πυρηνική ενέργεια. Αληθεύει αυτό. Τα ορυκτά καύσιμα όμως, πέρα από το ότι είναι πεπερασμένα και πέρα από το ότι έχουμε μεγάλη εξάρτηση από τρίτες χώρες μέσω αυτό, μειώνουν εκπέμπουν υψηλούς, ε, ε, υψηλές συμπυκνώσεις ε, ρήπων που επιβαρύνουν το περιβάλλον και έχουμε θέματα και με την πυρηνική ενέργεια αποβλήτων και θέματα ασφάλειας. Βλέπουμε λοιπόν ότι για το περιβάλλον αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Επίσης αληθεύει στον τομέα της έρευνας προχωράμε σημειώνουμε πρόοδο σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα για τη σύλληψη και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Σημειώνουμε πρόοδο σε σχέση με την έρευνα για πιο καθαρά καύσιμα και αληθεύει ότι και στην πυρηνική ενέργεια πάλι προχωρούμε όσον αφορά την αντιμετώπιση των αποβλήτων και την ασφάλεια των αντιδραστήρων. Έτσι λοιπόν σημειώνεται μεγάλη πρόοδος όσον αφορά και τις καθαρές πηγές ενέργειας, την καθαρή ενέργεια. Θα ήθελα να διαφοροποιήσω μεταξύ έρευνας και πολιτικής. Στην έρευνα πρέπει να είμαστε πολύ ανοιχτοί, να επενδύσουμε προς κάθε κατεύθυνση, διότι η ίδια ιστορία της επιστήμης μας δείχνει ότι δεν ξέρουμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθεί η σωστότερη λύση. Όμως από την άλλη μεριά στην ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να υπάρχει πολυμορφοποίηση και να υιοθετούμε το πιο ισορροπό ε, μείγμα, ενεργειακό μείγμα, σεβόμενοι το περιβάλλον και σε προσιτές τιμές. Για όλους αυτούς τους λόγους ποια θα ήταν η πρότασή μας. Λοιπόν, το ανέφεραν αυτό πιο πριν σύντροφοι που προηγήθηκαν και παρενέβησαν. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια εργαζόμαστε για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού. Είχαμε και το πρώτο πρόγραμμα δράσης 2007-2009 ε, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα αρμόδια κοινοτικά όργανα ήδη κάναμε μεγάλες προσπάθειες νομοθετικής ρύθμισης θέτοντας τα θεμέλια για τον ενεργειακό ανεφοδιασμό δρώντας ταυτόχρονα όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας μέχρι και την κατανάλωση. Και δράσαμε κυρίως επί τριών αξώνων, σε τρεις γραμμές, που θεωρώ ότι αυτές θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε στη δράση μας. Είναι η δημιουργία μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς με όλα όσα συνεπάγεται αυτό όσον αφορά δίκτυα και διασυνδέσεις και υποδομές μετά στη συνέχεια την ε, ε, ασφάλεια του ανεφοδιασμού να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά κατά τα τελευταία χρόνια και Καταρχήν αυτή θα ήταν η δική μου πρόταση, διότι θεωρώ ότι είναι η πιο σωστή πρόταση, η πιο σωστή πορεία. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχει το λόγο η κυρία Μαργκερίτα Μαστρομάουρο από την Ιταλία. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω μόνο να συμφωνήσω για την τελειώνοντας αυτή την ε, συνάντηση, ε, εκφράζοντας κάποιες ε, προβληματισμούς που προήλθαν από τις παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής της ομάδας εργασίας. Ένα από τα στοιχεία που προέκυψαν, σαφώς, είναι πως όλοι γνωρίζουμε τη σημασία μιας κοινή ενεργειακής πολιτικής. Ωστόσο, προέκυψαν και κάποιες βασικές διαφορές όσον αφορά τον αντοπισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων των χωρών, που όσον αφορά την επιλογή του ενεργειακού μείγματος, αλλά προέκυψε και κάποιο τύπος εγωισμού από πλευρά σε κάποιον πιο ανεξάρτητων χωρών από άποψη ε, από πλευρά των περισσότερων μου φαίνεται ότι οι περισσότεροι δεν συμφωνούν με τη δημιουργία μιας νέας ενεργειακής ε, συνθήκης και ο πρόεδρος Βόμποντα το επιβεβαίωσε αυτό. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή χρειάζεται συνεργασία στο θέμα και όχι κανόνες άλλους, αλλά συγκεκριμένες ενέργειες. Νομίζω πως όλα αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν μέσω των παρεμβάσεων και θα πρέπει με όλες οι χώρες να εκτιμήσουν, να κατανοήσουν το πλεονέκτημα του συνεργασίας μεταξύ τους και όχι να το δουν ως μια αύξηση των υποχρεώσεων. Νομίζω λοιπόν πως είναι πολύ σημαντικό και το είπαμε και στη γενικότερη συζήτηση, πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε και να ενισχυθούν οι επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές, τα κίνητρα για την ε, εξοικονόμηση ενέργειας και έπειτα πιστεύω πως είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιδέα μιας κοινή ε, προμήθεια, ενό κοινού ανεφοδιασμού μπορεί να δώσει πλεονεκτήματα και να προσφέρει καλές τιμές στις χώρες μέλη. Νομίζω πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να πείσουμε τα κράτη-μέλη να χάσουν λίγο από την κυριαρχία τους ένα στατηγικό τομέα για την οικονομία τους, εκτός αν όντως ε, τους δώσουμε μια ένα σαφές μήνυμα ευκαιρίες ε, και όχι υποχρεώσεων ακόμα και στο όνομα αυτής της ε, αρχής της ιερής που είναι η αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ντουκλάιφ Ιβανόφ από τη Βουλγαρία. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να πω, δίνοντας συνέχεια σε αυτά τα οποία είπε ο εκπρόσωπος της Σλοβακίας. Θα ήθελα να πω ότι αν υπάρχει μια χώρα που επλήγει τα μέγιστα από την κρίση του φυσικού αερίου, είπε, ήταν η Σλοβακία, όμως η δική μου χώρα επλήγει ακόμα περισσότερο. Είναι εκείνη που επλήγει χειρότερο από όλες τις άλλες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι Καμιά χώρα δεν έχει μεγαλύτερο συμφέρον και ενδιαφέρον στο να υπάρξει η ενεργειακή κοινότητα, ευρωπαϊκή ενεργειακή κοινότητα από ότι η Βουλγαρία. Οι ιδέες που εκφράσονται εδώ για την ενεργειακή κοινότητα της Ευρώπης και το ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ακούγονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά όλα, για όλα τα κράτη-μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Τρία σημεία θα ήθελα να θίξω, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ασφάλεια του ανεφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διασφαλιστεί με καλύτερο τρόπο μέσω της διασύνδεσης. Η δημιουργία αυτού του δικτύου διασύνδεσης θα δημιουργήσει την δυνατότητα για κάθε κράτος μέλος να έχει ένα, τη δυνατότητα παροχής ενεργειακών προϊόντων για τα ενεργειακά προϊόντα που χρειάζεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το φυσικό αέριο. Ένα άλλο σημείο το οποίο αναφέρθηκε και από τους προλαλήσαντες είναι η ανάγκη να βελτιώσουμε σημαντικά την ενεργειακή απόδοση και ε, τις ενεργειακές μας επιδόσεις και την αποδοτικότητα. Ως ένα μέλος του Συμφώνου της Βαρσοβίας στο παρελθόν ένα σημαντικό μέρος τμήμα της οικονομίας είναι ιδιαίτερα ε, ενεργοβόρο και η βελτίωση της αποδοτικότητας σημαίνει η διεύρυνση επέκταση φάλιας διότι θα έχουμε ανάγκη πρόσθετων ε, ενεργειακών προϊόντων. Όταν θα εξοικονομούμε όμως θα ε, μειώνεται η ανάγκη για αυτά τα προϊόντα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η πυρηνική ενέργεια είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, ενεργειακής πολιτικής στον 21ο αιώνα και ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά δημιουργεί, θέτει τρία ε, ζητήματα. Η δημιουργία νέων πυρηνικών αντιδραστήρων και σταθμών δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα έχουμε καλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Διότι στη Βουλγαρία βασιζόμαστε για το μεγαλύτερο τμήμα του ενεργειακού μας ανεφοδιασμού από μια χώρα, εξαρτώμαστε από μια χώρα. Το να δημιουργήσουμε ένα δεύτερο πυρηνικό αντιδραστήρα <clears throat> με βάση την τεχνολογία που παρέχει αυτή η ίδια χώρα με κανένα τρόπο δεν αυξάνει την ενεργειακή μας ασφάλεια. Και έτσι λοιπόν οδηγούμε στο τρίτο συμπέρασμα. Η πυρηνική ενέργεια ουσιαστικά βασίζεται σε ε, ένα ορυκτό καύσιμο, το ουράνιο. <clears throat> Και πρέπει εδώ να δούμε το θέμα του ουρανίου. Δεν είναι ίσως η πιο, ε, θα έλεγα, τα περισσότερα υποσχόμενα αυτό. Εν τέλει αντιμετωπίζουμε και το θέμα του τι συμβαίνει από πλευράς κάθε χώρας ε, όσον αφορά τα πυρηνικά απόβλητα. Τι συμβαίνει με τα απόβλητα. Όλες οι χώρες οι οποίες ε, αναπτύσσουν πυρηνικούς αντιδραστήρες πρέπει να δουν τη δυνατότητα εναπόθεσης και αποθήκευσης αυτών των πυρηνικών αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται ένα, καλό, ένα καλύτερο μέλλον για τις μελλοντικέ γενναίες. Διότι αν εξάγουμε τα πυρηνικά μας απόβλητα αλλού αυτό δημιουργεί την ίδια εξάρτηση όπως όταν κάποιος εξαρτάται από το πετρέλαιο. Διότι όταν ε, θέλουμε να εξάγουμε τα απόβλητά μας σε μια άλλη χώρα, αυτή η χώρα μπορεί να πει λυπούμαστε, δεν δεχόμαστε αυτά τα απόβλητα πια. My Έχουμε ακόμη δύο μιλητές. Οπότε θα έλεγα ε, μετά από αυτά τα δύο σχόλια να δώσουμε το λόγο στους συγητές γιατί έγιναν πολλές ερωτήσεις σήμερα και θα χρειαστούν χρόνο. Το λόγο έχει ο κύριος Γκάρτβολ από, το, από την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή και ο τελευταίος ο κύριος Σαρμπιζέ. Συμφωνείτε? Ωραία. Τότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκάρτβολ. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε εδώ βρίσκομαι και ζήτησα το λόγο. Ήθελα σαν εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με ορισμένες γνωμοδοτήσεις που έχουμε καταρτήσει. Διότι εδώ μιλάμε ουσιαστικά όταν μιλάμε για αντικατάσταση των ορυκτών πηγών ενεργείας, ε, για ανανεώσιμες και ορισμένες φορές και για πυρηνικές πηγές ενεργείας. Αλλά όλα αυτά είναι τεχνικές γιατί την παραγωγή ηλεκτρισμού. Ένα μεγάλο μέρος όμως αναγκών ε, ενεργεία στην Ευρώπη δεν ε, βασίζεται στον ηλεκτρικό τομέα όσο σημαντικός και να είναι αυτός αλλά και σε άλλους τομείς όπως η χημεία, ο άνθρακας, ιδίως οι μεταφορές, η θέρμανση και ούτω καθεξής. Γι' αυτό ήθελα πέραν της συζητήσεως για το πετρέλαιο και το αέριο να αναφέρω ότι ε, ε, η πηγή ενεργείας με τα μεγαλύτερα θέματα είναι ο άνθρακας ο οποίος βέβαια δημιουργεί και τα μεγαλύτερα ε, τη μεγαλύτερη παραγωγή ναι ναι ναι διοξιδίου του άνθρακος. Χρειάζεται λοιπόν ε, η τεχνική τη CCC, Carbon Capture and ε, Storage, Carbon Sequestration, ε, η οποία όμως έχει αμφιλεγόμενη αποδοτικότητα και εδώ έχουμε ένα δίλημα, διότι η τεχνολογία αυτή της δεσμεύσεως και της αποθήκευσης και του διοξιδίου του άνθρακος άνθρακα ε, σημαίνει ότι θα ε, καταναλώσουμε πιο γρήγορα το ακριβό αυτό υλικό από ότι αν το καταναλώνουμε κανονικά. Οπότε, εάν αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα απ' όλα είναι η επιδείνωση του κλίματος θα πρέπει ε, να πιούμε το μικρό ποτήρι να εφαρμόσουμε το CCS ε, για να μειώσουμε την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακος εάν όμως τα αποτελέσματα των ερευνών δεν επιβεβαιώνουν αυτό θα μπορέσει να μην εφαρμοστεί η τεχνολογία CCS αλλά ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν νέες τεχνολογίες αυτό ήθελα να επισημάνω και πάλι διότι εμφανίζεται ο άνθρακας σαν το, η ορυκτή πηγή ενεργείας η οποία έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα. Ευχαριστώ. Και ο τελευταίος ομιλητής που θα λάβει το λόγο απόψε είναι ο κύριος Μπισέ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε τελευταία φορά το λόγο διότι θέλω να τονίσω τον επίγοντα χαρακτήρα να ανταποκριθούμε στην πρόταση που μας έκανε ο κύριος Μπούζε και ο Ζακ Ντελόρ να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ε, ε, κοινότητα ενεργείας διότι υπάρχει μια πολιτική ε, πολιτικών που είναι μακριά στη διαρκείας και ε, πολιτική των ε, ε, επικεφαλής επιχειρήσεων ε, που είναι πιο βραχία. Ε, τώρα συνερχόμαστε από μία οικονομική κρίση τη χειρότερη από το κράχ του 29 και εδώ μιλάμε για τη στρατηγική του 2020 και νομίζω ότι θα ήταν αναχρονιστικό να μην εφαρμόσουμε αυτή την κοινή ενέργεια, ε, την κοινή ενεργειακή πολιτική ε, χωρίς να εφαρμόσουμε και την ενισχυμένη συνεργασία. Διότι εάν ορισμένοι ξεκινήσουν οι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε ε, την ε, επίρρεια εις την τιμή της ενεργείας η οποία θα πέσει και γι' αυτό μιλώ για οικονομία και για επίγουσα λήψη αποφάσεως η οποία επιβάλλεται. Ευχαριστώ κύριε και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον συγγητή μα, τον κύριο Σαρασβόλσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ποικιλία των θεμάτων που εφήγησαν στη συζήτηση δεν με επιτρέπει να αναφερθώ σε όλα όσα υπόθηκαν. Θα είμαι πολύ επιλεκτικός. Πρώτα απ' όλα θα αναφερθώ στον ομιλητή από τη Λιθουανία ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της εσωτερικής αγοράς. Καταρχάς, υπήρξαν κάποιες στιγμές στη συζήτηση που αναφέρθηκε η ενία αγορά που είναι ομάδα εργασίας 2 και το περιβάλλον που αφορά την ομάδα εργασίας 3. Τα αφήνω παράμερα αυτά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε θέματα ασφαλείας και ενιαία αγορά. Κανείς δεν αρνείται τη σημασία που έχει ενιαία αγορά της ενέργειας και όλοι παραδέχονται ότι είναι σημαντικό τμήμα της Ενία αγορά εν γέννη. Το, ερώτημα, το σχόλιο μου θα είναι και ερώτημα ταυτόχρονα. Μπορούμε να έχουμε ενιαία αγορά χωρίς ενιαία ασφάλεια. Μπορούμε να απελευθερώσουμε και να έχουμε πλήρως διαφανή ελεύθερη διακίνηση ενέργειας αν υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας όσον αφορά τον ενεργειακό φοδιασμό. Ρητορικό ερώτημα για να δείξω ότι αυτά είναι αλληλένδετα. Θα ήθελα να αναφερθώ στο Λόδο Λόπερ, ο οποίος έθεσε κάποιο ερώτημα. Τι με εξέπληξε σε αυτά που είπατε. Είπατε ότι η Βρετανία δίσταζε να αναφερθεί στην ασφάλεια της ενέργειας και τώρα που βλέπει το τέλος των αποθεμάτων στη Βόρεια Θάλασσα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, η Βρετανία είναι πιο έτοιμη να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ο Τσάρλ Τάνοκ είναι εκεί. Θυμάσαι, Τσάρλ, πόσο δύσκολο ήταν να πείσουμε του Βρετανού συναδέλφους ότι χρειαζόμαστε σε αυτό το τομέα. Το σχόλιο μου θα ήταν ότι σήμερα, μάλλον χτε ήσασταν πλούσιοι σε φυσικό αέριο και αύριο θα είστε φτωχοί. Και χώρε οι οποίε είναι πλούσιε και αύριο θα είναι φτωχέ. Αλλάζει το ενεργειακό τοπίο. Ε, διότι δεκαετίε έτσι θα προχωρήσουν και θα κυλήσουν. Άρα αυτό μας δείχνει ότι χρειαζόμαστε κοινή προσέγγιση και όχι ατομικιστική, εγωκεντρική. Ε, δεν χρησιμοποιήθηκε η λέξη εγωιστική, αλλά για να το πούμε ομά. Μιλάμε για εγωκεντρική προσέγγιση. Μιλάμε για εγωισμό ή ελληνική. Για τα τρία ερωτήματα του Λόρδου Λόπερ, λοιπόν. Ή ρωτήσατε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει κάτι. Ναι, υπάρχει μια στρατηγική. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει έλλειψη προθυμία για να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Και ο περίφημο κανονισμός για το φυσικό αέριο που αναφέρθηκε επανειλημμένα που ουσιαστικά αποτελεί ορίμαση το άρθρου 100, υλοποίηση μάλλον του άρθρου 194. Το πρώτο κείμενο το αρχικό ήταν φιλόδοξο. Μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε με τα κράτη-μέλη και κατέληξε στο να παράγει κάτι που είναι άκρος μη φιλόδοξο. Και μετά τη συζητήσει στο Συμβούλιο το τελικό κείμενο ήταν ακόμα λιγότερο φιλόδοξο. Προσπαθήσαμε τώρα να το κάνουμε ξανά φιλόδοξο. Και δεν θέλω να προβώ σε προβλέψεις, αλλά κινδυνεύουμε να αποτύχουμε. Ένα πρόγραμμα πολύ φιλόδοξο πολιτική βούληση του Κοινοβουλίου θα ξεψυχήσει λόγω ελλείψεως ενθουσιασμού, για να το πω εφημιστικά, από πλευρά των κρατών μελών. Μακροπρόθεσμη στρατηγική, σαν έννοια ναι. Θα επιβιώσει όμως. Φοβούμε ότι ίσω όχι. Αν ε, δεν δημιουργήσουμε επαρκή πολιτική βούληση. Αναφερθήκατε στα αποθέματα πετρελαίου, είναι 90 ημέρες. Ασφάλεια, βιωσιμότητα, χρησιμο... χρειαζόμαστε άλλες δύο να συζητήσουμε αυτά. Και τέλος, στο φίλο μας Λεκεγέ που δεν είναι στην αίθουσα όμως αν δεν κάνω λάθος. Θα συνεχίσω αγγλιστή λοιπόν, εν τη απουσία του. Αναφέρθηκε και στη Ρωσία, θα σε ερώτημα για τη Ρωσία. Εμείς από τις χώρες της κεντρικής καθολικής ε, ε, Ευρώπης έχουμε βαρεθεί να λέμε που προέρχεται η ε, απειλή. Είναι καλό να τα ακούμε από το Παρίσι καμιά φορά. Αν δείτε τι έγινε στην Ουκρανία και τι συμβαίνει στη Λευκορωσία χάνουμε τη γειτονιά μας διότι η ενέργεια χρησιμοποιείται ως πολιτικό όπλο. Είναι ξεκάθαρο. Ακόμα και η παράταση της παραμονής του ρωσικού στόλου στη Σεβαστόπολη και το, η πίεση που κατά του Λουκασένκο. Ναι, τα έχουμε υπόψη αυτά και λεκυγέ. με την άποψή του ότι το μέλλον είναι η πυρηνική ενέργεια καποια κάτι κράτη-μέλη δεν τη θέλουν, αλλά ξέρω ότι οι Γερμανοί είναι πολύ διστακτικοί. Αγοράζουν πρόθυμα την ηλεκτρική σας ενέργεια που παράγεται από τους πυρηνικούς σταθμούς και μετά δεν έχουν δισταγμούς δεντολογικούς ή πράσινους δισταγμούς να αγοράσουν. Έχουμε όλα αυτά τα μείγματα τα ενεργειακά ή σημείο αυτό που είπατε. Το μπουκέ ενεργετικό αυτό ενεργειακό μπουκέτο με διαφορετικά ενεργειακά μπουκέτα μπορούμε να είμαστε πλέον συμπληρωματικοί όσον αφορά τα διαφορετικα κρατη κράτη-μέλη. Τώρα στον κύριο Λεκυγέ επιστρέφω. Συμφωνώ μαζί του ότι η πολιτική βούληση είναι το βασικό έλλειμμα έγκυται εκεί, βασικό θέμα αυτό. Πιστεύω, όπως πιστεύετε και εσείς, ότι θα πρέπει να δοκιμαστεί ένα μοντέλο τύπου Σέγγεν, ενισχυμένη συνεργασία ο μόνος φόβος μου είναι ότι θα έχουμε σύγκρουση μεταξύ φτωχών και εκείνων που έχουν ανάγκη. Εκείνοι που έχουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο θα μαζευτούν, αλλά δεν θα παράγουν πλούτο φυσικού αέριου. Και κάποιες, μάλλον οι χώρες που δεν θέλουν αλληλεγγύη, χωρίς να τις αναφέρω, είναι αυτές που τα καταφέρουν μια χαρά. Έχουν πόρους ή που ήταν πολύ έξυπνες εδώ και πολλά χρόνια, χάρη σε κάποιες ιδέες του στρατηγού De Gaulle, δεν αναφέρω προφανώς τη χώρα στην οποία αναφέρομαι, που επένδυσαν στον πυρηνικό τομέα, που τώρα είναι η ευλογία του Θεού για τη χώρα. Ή άλλους πολύ καλά ενεργειακά με διάφορους αγωγούς, με άλλες υπήρους, ας το θέσω έτσι. Καλή ιδέα αλλά αν δεν έχουμε εκείνους που θα μπορούσαν να προμηθεύουν στην αλληλεγγύη και μόνο εκείνους, έχουμε μόνο αυτούς που χρειάζονται τον εφοδιασμό από πλευράς αλληλεγγύης, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Ακούστηκαν φωνές πολλές. Κάνουμε διάκριση όμως μεταξύ μακροχρόνιας ασφαλείας, έρευνα, ανανεώσιμες, νέες πηγές και το καθεξής και των άλλων. Είναι διαφορετικό αυτό, είναι στρατηγική, δεν είναι ασφάλεια στατική για 20-30 χρόνια. Ασφάλεια είναι βραχυπρόθεσμη. Ο Σλοβάκο ή ο Βούλαρο συνάδελφου θα είπε ότι λύψει το αέριο τη χώρε, όταν σταματήσουν δημόσιο μεταφορέ, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τεργοστάσια λόγω λήψη φυσικού αερίου, απειλή που συγκρίνεται με εμπόλεμη κατάσταση, με βαμβαδισμό. Μπορεί να παραλύσει η χώρα χρησιμοποιώντας αυτό το ειπε οταν λειψει το αεριο απο τι χωρε οταν σταματησουν δημοσιες μεταφορες τα νοσοκομεια τα σχολεια τα εργοστασια λογω ελλειψεω φυσικου αεριου απειλη που συγκρινεται με εμπολεμη κατασταση με βομβαρδισμο μπορει να παραλυσει η χωρα χρησιμοποιωντα αυτο το οπλο Βραχυπρόθεσμη λοιπόν είναι η ασφάλεια. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο. Λιγότερο πετρέλαιο, διότι είναι εμπορεύσιμο να το αγοράσει κανεί στην αγορά Spot στο Ρότερνταμ. Αλλά υπάρχουν οι πιέσει όσον αφορά την ασφάλεια στο φυσικό αέριο. Όπω προανέφερα όμω, συμφωνώ με το Λεκυγέ. Έχουμε γεωπολιτικέ συνέπειε. Είμαστε εν το μέσο του να απολέσουμε τους ανατολικούς γειτονές μας λόγω τη χρήση αυτού του μέσου. Και αν κάποιος ήταν αρκετά έξυπνος να τραβήξει την, τη γραμμή μεταξύ δίκτου δημοκρατίας και δίκτου τιμής του φυσικού αερίου, βλέπεις όσο πιο δημοκράτης είσαι, τόσο πιο ψηλό το τίμημα που καταβάλεις και τούμπαλιν. Είναι γεωπολιτικό μέσο. Δεν είναι εμπορεύσιμο αγαθό. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον στα πλαίσια σημερινή κρίσεως και δεν συμφωνώ με κάποιον που είπε ότι πέρασε η κρίση. Είμαστε στο δεύτερο κύμα και κάποιες, κάποιοι οικονομολόγοι λένε ότι μας περιμένει και τρίτο κύμα. Το δεύτερο κύμα συμβολίζεται από την Ελλάδα. Αλλά δεν έλειξε το πρόβλημα. Δεν θα μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση αν δεν έχουμε φυσικό αέριο, αν δεν έχουμε ενέργεια σε προσιτέ τιμέ και αν έχουμε μονοπολιστικού προμηθευτέ στι αραβικέ χώρε και στη Ρωσία στο πετρέλαιο μονοπόλιο στο φυσικό αέριο, σε αυτή την προμήθεια. Και οι προσπάθειε οι ανησυχητικέ να δημιουργηθεί ο πεκ φυσικού αερίου. Και κοίτα τώρα, με την παραγωγή του φυσικού αερίου από διάφορα είδη άμμου στην Αμερική βλέπετε για χίλια κυβικά πληρώνω 300 δολάρια από τη Ρωσία και τιμή σποτ στο Ρότερνταμ υγροποιημένου αερίου είναι 150 τι σημαίνει αυτό, ότι πληρώνουμε δύο φορές για το ρωσικό αέριο από ό,τι θα έπρεπε. Και αυτό υπονομεύει τις απασχόληση, απασχόλησης, μειώνει του ρυθμούς ανάπτυξης και υπονομεύει την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης. Κάποιο είπε, ρώτησε ποιο θα τα πληρώσει όλα αυτά, Κύριο Βίτροτ Και τι χρειαζόμαστε όσον αφορά τι ε, κρατικές Όποτε αποτυγχάνει μια αγορά, ένα κράτο μέλο αποτυγχάνει και έχει προβλήματα, θα πρέπει να παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν δημόσια αρχή και σαν χρήματα. Διασυνδέσει που δεν είναι βιώσιμε οικονομικά θα πρέπει να καλύπτονται από τον κοινό μα προπολογισμό. Εάν πρέπει να δημιουργήσουμε αποθέματα, εκείνοι που επενδύουν θα πρέπει να απαριθμούνται και η πρόταση του κειμένου κανονισμού έλεγε ότι θα πρέπει να αμείβονται για τις επενδύσεις τους. Αν κάποιος κατασκευάσει υποδομές και αποθέματα θα πρέπει να αμείβεται. Αναλόγως. Χρειάζεται λοιπόν κάποια ασφαλιστική πολιτική που θα εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, στο ερώτημα Χρειαζόμαστε 20, με 27 πολιτικών ή κοινή πολιτική όσον αφορά αυτό το θέμα. Απαντώντας στον κ. Βίτπροντ λέω, ναι έχουμε ένα όραμα. Αλλά δεν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση. Ποιος θα πρέπει να πληρώνει ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ναι, απάντησα. Για να παριθμίσω τις προσπάθειες επενδυτικές, κύριε Μπιζή για τα κράτη-μέλη, και επιχειρήσει που να έχουν κίνητρα για να επενδύουν στην αποθήκευση, στις υποδομές κλπ. κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες αγοράς. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να παρεμβαίνουν όταν η αγορά δεν λειτουργεί πλέον. Για τον Αμπούκο και αναφέρομαι στον Τούρκο συνάδελφο περιπλοκότατο θέμα. Δεν θα είναι θάρρυνα τους Τούρκους φίλους μας να συνδέουν τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη με την συμμετοχή και την αλληλεγγύη με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Διότι αυτό μπορεί να παρεξηγηθεί. Ξέρω ότι έχει προβλήμα η Τουρκία με τι διαπραγματεύσει. Είναι οδυνηρέ διαπραγματεύσει. Το να χρησιμοποιείτε την, τα θέματα ενεργειακή ασφάλεια έτσι ε, δεν εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα. Κλείνοντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα όραμα, έχει φιλόδοξο πρόγραμμα, φιλόδοξα προγράμματα. Υπάρχει σαφή κίνδυνο αποτυχίας. Το λέω ξεκάθαρα αυτό. Κα, καλές ευχές, έξοχες παρόλα αυτά είμαστε κοντά στο να χάσουμε τη μάχη. Και με αυτόν τον ενσυχητικό τόνο θα κλείσω την παρέμβασή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σάρος Βόλσκι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Πρέπει να πω ότι με τιμά το ότι μπόρεσα να συμπροεδρεύσω αυτή τη σου απόψε. Όπως είπατε πολύ από σας, αν τα κράτη-μέλη κινηθήκαμε ατομικιστικά και όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια. Η Σουηδία σε 10 μέρες θα ψηφίσει στο Κοινοβούλιο και εκεί θα δούμε κατά πόσο και εμείς θα ακολουθήσουμε νέο δρόμο όσον αφορά την ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας. Θα επηρεάσει πολύ τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ενέργεια στη Σουηδία, στο μακρινό μέλλον. Προσβλέπω σας ξαναδώ και μεγάλη μου χαρά που άκουσα όλα τα όμορφα επιχειρήματά σας και θα πάρω μαζί με αυτά τα επιχειρήματα για να τα προβάλλω, να τα χρησιμοποιήσω συζητήσεις που ακολουθήσουν για την ενέργεια στη Σουηδία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.